Δεν μπορώ να περιμένω περισσότερο γιατί έχουμε πάρα πολλά θέματα να συζητήσουμε αλλά θα πρέπει επίσης να σας ενημερώσω για τις χθεσινές ε, αποφάσεις των συντονιστών και που θα πρέπει να τις ε, εγκρίνουμε. Αποφασίσαμε σε σχέση με την ε, διάθεση των πόντων σε ομάδες και βουλευτές. Και οι συντονιστές είπαν ότι 7 θα πάνε σε κάθε βουλευτή σε κάθε πολιτική ομάδα. Και επίση θα ισχύσει το ίδιο σύστημα διάθεση εκείνο το οποίο ανέκαθεν ίσχυε. Δεύτερον, όσον αφορά την ε, διάθεση και ορισμό ε, συντακτών γνωμοδοτήσεων, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοκράτε όσον αφορά το νομοθετικό έργο και όσον αφορά τις νομοθετικές γνωμοδοτήσεις, και εκθέσεις. Το πρόγραμμα για καινοτομία και έρευνα θα το πάρει το ECR ε, για το Ταμείο την Αλία το ΕΛΚ, για το περιβάλλον, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες και τώρα σε σχέση με τον οργανισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το στατιστικό πρόγραμμα 2017 Αυτό θα εκκρεμεί για μία εβδομάδα. Δεν ελήφθη καμία απόφαση όσον αφορά την οδηγία για κάποιες συμβάσεις η πράσινη οδηγία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για δημόσιες προμήθειες η Άλντε. Η Άλντε επίσης και την άλλη οδηγία για τις ε, προμήθειες για ταχυδρομικά ύδατα Τώρα όσον αφορά το προενταξιακό μέσο βοήθειας το ΕΛΚ, ε, μέσω γειτονίας ε, πολιτική γειτονία, το ΕΛΚ, δημογραφία, σοσιαλιστές, μηχανισμός ε, πολιτικής προστασίας, ECR. Μη νομοθετικές νομοθετήσεις, δύο αποφάσεις ελήφθησαν όσον αφορά τα καινοτόμα μέσα για το MFF, οι σοσιαλιστές για το πολιτές πλαίσιο, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Άλντε. Και επίσης οι συντονιστές συμφώνησαν να ενημερωθεί η γραμματεία το νωρίτερο δυνατόν όσον αφορά τις προτιμήσεις, όσον αφορά τον αριθμό των μελών που θα λάβουν μέρος στις τρεις ε, αντιπροσωπείες που αποφασίστηκε σε κάποια φάση να γίνει τέτοια ενημέρωση το νωρίτερο δυνατόν. Επίσης συμφωνήθηκε ότι όταν πάμε στην Κόπενχάγη δεν θα αφορά μόνο συνάντηση με την Προεδρία. Θα ασχοληθούμε με θέματα ευρύτερα. Α, θα δούμε. Ο κ. Φανίστελ Ρόε ζήτησε από την ε, γραμματεία να γίνει μια εισήγηση για την κατάσταση των πραγμάτων για το κατά πόσον τώρα μπορούμε να έχουμε εκθέσεις ιδίας Πρωτοβουλία. Και θα συνεχίσουμε τις επαφές, επί συζήτηση ο κ. του ΛΟΕ, η Γραμματεία, να συνοθεί με την Ήτρεμ πως μπορούμε να έχουμε κοινή ακρόση όσον αφορά την κλίμακα αριστείας. Το Μάρτιο επίσης να δούμε τι θα γίνει με κάποια παρουσίαση μελέτης για την πολιτική, ε, για τα πολιτιστικά στην Αυστρία. Όλα αυτά τα απεφάσισαν οι συντονιστές. Όλα αυτά είναι οι προτάσεις προς την Επιτροπή. Τώρα, Πάμε στο σημείο 18, πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα θέματα που παραδοσιακά παρουσιάζουν δυσκολίες όσον αφορά τη σχέση του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου και των πολιτικών μας. Ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τους ε, εισηγητές του προϋπολογισμού έχουμε και εκπροσώπους της Επιτροπής των Περιφερειών. Επίσης, δεν μπόρεσαν να παραστούν στη συζήτησή μας ούτε ο ένας ούτε ο άλλος από τους ε, εισηγητές του προϋπολογισμού. Συνέφεξε το λόγο. Μεγάλη μου χαρά τώρα να σας παρουσιάσω αυτό το έγγραφο που αφορά το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 14-20 καθώς και τις επιπτώσεις επί της συνοχής. Πρώτα πρώτα όσον αφορά τη διαδικασία συζητούμε μόνο τα βασικά, τις βασικές αρχές σε σχέση με τη διάθεση των πόρων την περίοδο αυτή. Οπότε να δούμε τι γίνονται τα αριθμητικά στοιχεία σε επίπεδο των μελών. Έχουμε την ε, εντολή του Συμβουλίου προς την ε, Προεδρία. Και αυτό θα γίνει τον Ιούνιο. Προτείνεται αυτό το πλαίσιο με στόχους την απλούστευση της εκτονικής των πολιτικών. Απασχόληση, ανάπτυξη και ανάπτυξη της πέθρου. Αυτό είναι ένα κλάσμα των χρημάτων που θα δοθούν στην πολιτική συνοχή. Πρέπει όμως να μην ξεχνούμε ότι θα γίνει διαβούλευση από πάνω προς τα κάτω και ενδεχομένως υπάρξουν περαιτέρω περικοπές των ποσών που προβλέπεται αρχικά να διατεθούν. Κάποιες παρατηρήσει μου πρώτα-πρώτα για το 2,5% του ΕΠ όπως καθορίστηκε Και έχουμε εδώ πέρα μια αναθεωρημένη εκδοχή του εγγράφου, γιατί ε, σε σχέση με το. Σε αρχή είχαν πει GNI, ότι 2,5% αλλά δεν είναι του GNA είναι του GDP, του ΑΕΠ δηλαδή ο υπολογισμό αυτό. Όσον αφορά αυτά τα άνω όρια των μελών, πάμε λοιπόν για το όριο του 2,5%. Εγώ δεν ξέρω ότι αυτό δικαιολογείται και θα είναι πάρα πολύ ανεπαρκέ για κάποιε περιφερειέ όσον αφορά την πολιτική τη συνοχή. Για μένα επομένω, αυτό το ποσοστό δεν είναι το πιο σωστό και ώρα να προχωρήσουμε σε ανταλλαγή απόψεων για να δούμε τι θέση θα αποκρισταλώσουμε. Το ποσοστό αυτό αφορά κάποιες περιφέρειες. Θα πρέπει επίσης να προσεχθούν όσο αφορά την κάλυψή τους για την επόμενη ε, δημοσιονομική χρήση. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι θα ισχύσει η ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των κανόνων. Ε, αυτά που είπαμε και χθε τα βόηματα θα τα πούμε και προκειμένου όσον αφορά την ε, απόδοση της επιδόσεις ε, και την ανταμοιβή προς τις πιο αποδοτικές περιφέρειες. Άρα θα πρέπει οι περιφέρειες να ορίσουν στόχους που να μην είναι τόσο φιλόδοξοι που μπορούν να τους πιάσουν. Και αντιστοίχω οι χώρες να μπορούν να απορροφήσουν αυτό που τους διατίθενται. Άρα, θα πρέπει το σχετικό αποθεματικό θα πρέπει να οριστεί σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, το επόμενο σημαντικό θέμα το οποίο και αυτό συζητήθηκε χθε είναι η αυτόματη συγκέντρωση. Εδώ σαφώς χρειάζεται ευελιξία. Και διαπιστώνουμε ότι από τη μια μεριά είναι θετικό το να υπάρχει ευελιξία, το πολιτικές πλαίσιο θα πρέπει να τα πάει καλύτερα από ότι η πορεία για τη συνέχεια της Λισαγώνας όσον αφορά τους στόχους που τίθενται όμως υπάρχει πολυμορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να γίνει ενιαία αντιμετώπιση. Άλλο βορρά, άλλο νότο, ανατολή, δύση. Άρα εδώ πέρα θα πρέπει να διευνήσουμε τη δυνατότητα μήπω μπορούν οι περιφέρειες να έχουν διακριτική ευχέρεια να επιλέξουν την μορφή, την εκδοχή ευελιξία. Τώρα όσον αφορά την ποσόστοση, το ποσοστό, όπως θέλετε πέστε το, τρεις κατηγορίες περιφερειών μπορούμε να πούμε ότι προβλέπονται. Νομίζω ότι το ποσοστό αυτό είναι υπερβολικά φιλόδοξο, όπως το λέει η Κομισιόν. για τις προτεραιότητες 80, 60 και 50 Ιδίω για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες θα πρέπει να πάμε πιο χαμηλά να έχουμε πιο χαμηλά τον πύχη για τις δαπάνες υποχρεωτικής συγκέντρωσης. Παρακαλώ, με ενδιαφέρει πάρα πολύ να πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτά. Είπαμε ε, ότι εδώ πέρα στοχεύει η Κομισιόν σε αυτές που, είναι, ε, που έχουν ΑΕΠ κάτω από το 90% του μέσου όρου. Και έχουμε εδώ κάποια έργα υποδομών, προγράμματα αντίστοιχα, όμως αυτό το οποία εδώ προβλέπονται είναι κάπως ε, ασαφή, χρειάζεται περισσότερη διασάφηση, ε, πώς θα γίνεται η επιλογή, πώς θα γίνεται η διαχείριση κλπ. 5% του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης θα πέσει κάποιες ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη των ε, πόλεων και αυτό το θεωρούμε θετικό. Να δούμε πώς θα ξεκαθαριστεί η πρικοδότηση του κοινωνικού ταμείου. Να δούμε πώς θα είναι πιο αποτελεσματικές ταπάνες για τους ανθρώπινους πόρους. Σας υπενθυμίζω επίση ότι υπάρχει κάτι σημαντικό διαδικαστικό σύμφωνα με το άρθρο 312 της συνθήκης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να πει ναι ή όχι. Και τίποτα άλλο όσον αφορά το πολιετές πλαίσιο. Όμως, το άρθρο 1 του κανονισμού μας λέει ότι η αρμόδια επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παρουσιάσει ενδιάμεση έκθεση για το πολιετές πλαίσιο και ψήφισμα με συστάσεις για τροποποίηση και εφαρμογή της πρότασης. Η δημοτευτική εντολή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν το τέλος της Προεδρίας. Όμως ε, η Επιτροπή των Προπολογισμών ακόμα δεν αποφάσισε για την έκθεση. Όπως και έχουν τα πράγματα, αυτό δεν μας ε, αποκλεί το να προχωρήσουμε εμείς προς αυτή την έκθεση για την πολιτική της συνοχή και τη συνέπειες. Περιμένω πώ και πώ να ακούσω την άποψή σα σήμερα. Συνάδελφοι, να ανταλλάξουμε απόψει, να ακούσω και τι έχει να πει και η Επιτροπή των Περιφερειών. Δυστυχώ, δεν έχουμε εδώ του συζητητέ των προπολογισμών. Να μα πούνε πώ έχουν εκεί τα πράγματα. Ελπίζω και με αυτού να έχω αγαστή συνεργασία και σίγουρα να έχω και αγαστή συνεργασία και με την Επιτροπή των Περιφερειών. Ε, πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ. Οι τώρα. Ο Γιώργος Αβρακάκης, της πρώτος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το έγγραφο εργασίας που μόλις παρουσίασε και για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει. Ε, οι δύο εισηγητέ μα για το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο διεξάγουν τι διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο με βάση την ξεκάθαρη εντολή που του έχει δοθεί από την έκθεση τη Ειδική Επιτροπή ΣΥΟΡΕ στην οποία αρκετοί από εμά ήμασταν μέλη και η οποία διαθέτει ένα ειδικό κεφάλαιο για τα θέματα τη πολιτική συνοχή. Συμφωνώ με την ανάλυση του εισηγητή και την υποστηρίζω εκτός από το τελευταίο σημείο που αναφέρεται στα υποχρεωτικά ποσοστά του Κοινωνικού Ταμείου. Είναι πάγια η θέση της Επιτροπής μας, όπως παρουσιάστηκε και χθες από τους δύο εισηγητές του Γενικού Κανονισμού, ενάντια στην υποχρεωτική χρήση ποσοστών μια και λειτουργεί ανασταλτικά στη δημιουργία χάραξη πολιτικών ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περιφέρειας prevent needs based policy making. Θα σταματήσω εδώ μια και συμφωνώ με τα υπόλοιπα σημεία του εγγράφου του συγητή και να τον ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά για την πολύ καλή δουλειά που ε, μας παρουσίασε. Mm. Με συγχωρείτε, ε, ο κύριος Τόιρερ νομίζω ότι δεν είναι εδώ, οπότε θα ήθελα να ρωτήσω ποιος ε, άλλος θέλει να ε, τον αντικαταστήσει. Η ομάδα μας για το έχει αρκετά ευθυγραμμισμένες θέσεις με την Επιτροπή Προϋπολογισμού σχετικά με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Δηλαδή θέλουμε να διαφυλάξουμε μια πολιτική, ε, περιφερειακή πολιτική μέσα στο πολιετές πλαίσιο και πρέπει εμείς να παράσχουμε όλα τα σχετικά επιχειρήματα. Διότι η περιφερειακή πολιτική αποτελεί πραγματική υπεραξία στην Ευρώπη για να καταπολεμήσουμε την κρίση και να βοηθήσουμε τις ε, περιφέρειές μας να αντιμετωπίσουν ε, την κρίση. Πρόκειται για την πραγματική ευρωπαϊκή σφραγίδα. Και το να κάνουμε περικοπές στην περιφερειακή πολιτική είναι σαν να εναντιονόμαστε στην ίδια την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή ιδέα. Τώρα, η Επιτροπή έχει συγκεκριμένους ε, στόχους και ένα πλαίσιο που δεν είναι ιδιαίτερα ευέλικτο στις προτάσεις ε, που, που κάνει. Αυτό το οποίο λείπει σήμερα από την Κομισιόν ε, είναι μία πρόταση που δεν είναι ευέλικτη, δηλαδή μία πρόταση μονόδρομος. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι θέσει των περιφερειών στον μελλοντικό προγραμματισμό. Θα πρέπει να υπάρχει ένας πραγματικός μηχανισμός διαπραγμάτευσης και ανταλλαγών ούτως ώστε ο κάθε τοπικός παράγοντας να μπορεί να έρχεται με τις προτεραιότητες του, να έρχεται και η Ευρώπη με τις δικές της προτεραιότητες και να υπάρχει μια μεγαλύτερη διαβούλευση τη στιγμή της αλήθειας. Το διάβημα σήμερα το οποίο ξεκινάμε είναι τεράστιες αξίας για την Ευρώπη. Ευχαριστώ Φρανσουά. Τώρα θα έλεγα να ε, συζητήσουμε και να ακούσουμε τον Φλοκ που είναι ο, ο εισηγητής. Ή Κλοντ, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι που μου δίνετε το λόγο. Άκουσα αυτά που είπαν οι συνάδελφοι και ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε ε, ε, αυτά που λέμε και εμείς ε, στην γνωμοδότησή μας που στηρίζει την εργασία των συναδελφών σήμερα διότι οθετήσαμε την γνωμοδότηση αυτή και πρέπει να πω με περηφάνεια για το Ηνωμένο Βασίλειο ότι κανείς δεν την καταψήφισε παρόλο που αναφέρεται στον φόρο δημοσιονομικών ε, ε, ε, οικονομικών συναλλαγών και είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι. Θεωρούμε ότι αυτό είναι το σημείο που ξεκινάμε για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις διαπραγματεύσεις και υπάρχουν και διάφοροι στόχοι πολιτικοί σε αυτό τον χώρο. Καταρχήν θέλουμε να στηρίξουμε την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθούν μεταβατικές περιοχές και ήδη οι πόροι και επιπλέον ε, θέλαμε να ε, ε, στηρίξουμε και την αιρεσιμότητα που είναι πολύ σημαντική διότι είναι προφανές ότι ο λόγος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή την περίοδο έχει ενισχυθεί και θα θέλαμε να υπάρχει πλήρη συναπόφαση με τους άλλους που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες και πιστεύουμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρτήσαμε την πρόταση ε, προσπαθώντας να εμπλέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ενδιαφερόμενους και εδώ αναφέρομαι στο Ευρωπαϊκό ε, Κέντρο Πολιτικής, σε ε, ε, ε, δημιουργήσαμε διάφορα εργαστήρια με όλους ε, τους ενδιαφερομένους και από το σχετικό χώρο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολιτικές ομάδες και εθνικές αντιπροσωπείες και θέλαμε να τους ενημερώσουμε τι λέει ε, η Επιτροπή Περιφερειών επ' αυτού διότι πιστεύω ότι αυτοί είναι άμεσα εμπλεκόμενοι και πρέπει να μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους για να ε, μπορέσουν να στηρίξουν αυτά τα οποία ε, επεξεργάζεται η Επιτροπή σας. Αυτά όσον αφορά τη γνωμοδότηση την οποία συνδυάζουμε με την πολιτική συνοχή. Όσον αφορά την δομή του προπολογισμού πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες που έχουν διατυπώσει τα κράτη-μέλη στην ατζέντα του 2020. Δεν είναι δυνατόν να λέει κανείς ε, ε, μία άποψη στις Βρυξέλλες και τελείως το αντίθετο όταν απομακρύνεται. Και ε, πιστεύουμε ότι ο στόχος είναι να υπάρξει ένα πλήρες πρόγραμμα διαρθρωτικό το οποίο να συνάδει με τον παρόντα γύρο των διαβουλεύσεων κατά τρόπον ώστε να υπάρξει συνοχή η οποία θα μπορέσει να υλοποιήσει το πρώτο κεφάλαιο του προπολογισμού διότι ε, σύμφωνα με αυτά που έχουμε συμφωνήσει δεν θα μπορεί πλέον να μεταφέρει ε, κανείς τα χρήματα που δεν έχουν δαπανηθεί σε ένα άλλο σημείο και αυτό θα το συζητήσουμε. Ε, ε, ε, επίσης είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη αιρεσιμότητα που θα ήταν αντιπαραγωγική για να μπορούμε να υποκινήσουμε τις περιφέρειες να ξοδέψουν αυτά που περιέχει ο φάκελος συνοχής. Πρέπει επίσης να υπάρχει συνεκτικότητα των προγραμμάτων, να εμπλακούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και όχι απλώς να εφαρμόζουμε την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής ε, Ενώσεως. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης σχέση συνεργασίας και ε, ε, επαναλαμβάνω την άποψη της Επιτροπής ε, Περιφερειών η οποία πιστεύει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αποθέματα τα οποία θα βασίζονται σε προσυμπεφωνημένους εθνικούς φακέλους παρά μόνο υπό ειδικέ προϋποθέσεις. Δηλαδή εάν ε, δεν υπάρχει υλοποίηση των αποτελεσμάτων που στα οποία προβλέπει κανείς και θέλουμε ε, συγχρόνως να αποφύγουμε η ε, διακοπή παροχής ε, ενισχύσεως ε, να γίνεται αυθαίρετα και όχι βάση μέτρων. Είμαστε αντίθετοι ότι, στο ότι πόροι ε, θα πρέπει να, ε, ε, βασίζονται σε μεμονωμένες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να ικανοποιήσει κανείς τις περιφέρειες και να τις βοηθήσει να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και θα πρέπει να υπάρχει η ισότητα των φύλων, δεύτερον ο πολιτισμός να αποτελέσει το μέσο για να αναπτυχθούμε και ε, να βοηθήσουμε την επιχειρηματικότητα ιδίως των νέων οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν στις περιφέρειές τους. Όσον αφορά τον στρατηγικό προγραμματισμό θεωρούμε ότι το Ταμείο θα πρέπει να παραμείνει εδρεωμένο ή στην ευρωπαϊκή πολιτική και να υπάρχει ένα ενιαίο σύστημα κατευθυντηρίων γραμμών βάσει των αρχών που προενέφερα. Από πλευράς στρατηγικής πιστεύουμε ότι περισσότεροι πόροι πρέπει να πηγαίνουν εις τις πιο φτωχές περιοχές για να μπορέσουν να ανταποκριθούν εις τις προκλήσεις διότι υπάρχουν περιοχές στις κοινότητές μας παντού που δεν πρέπει να αποκλειστούν διότι δεν έχουν τους αναγκαίους ιδίους πόρους πρέπει να υπάρχει δε μία νέα μεταβατική κατηγορία περιοχών και δεδομένου του ότι είπε ο κύριος Κόβατσεφ ήδη θεωρούμε ότι ε, δεδομένου στις αφομοιώσεις το πλαφόν δεν θα πρέπει ε, να, ε, να παραμείνει στα επίπεδα της περίοδου που έχουν καταρτιστεί για τα κράτη-μέλη για την περίοδο 2007-2013 διότι θα ήταν εις βάρος όλων. Θα πρέπει η τοπική αυτοδιοίκηση να θεωρηθεί ισότιμος εταίρος και να υπάρξουν συμφωνίες ε, συνεταιριστικές ε, και να μπορούν ε, να δημιουργηθούν ε, ε, συνεργασίες με τις εθνικές κυβερνήσεις η δε τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να επιτηρεί τα προγράμματα τα οποία καταρτίζονται δεν υπάρχει κανένας λόγος να υπάρχει διαχείριση ενός προγράμματος σε μία περιοχή αν δεν συμμετέχει η τοπική αυτοδιοίκηση της περιοχής περιοχής. Και τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω διότι πολλοί συνάδελφοι μπόρεσαν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία και ε, να σας πω ότι ε, μόνο δύο συνάδελφοι από το Ηνωμένο Βασίλειο καταψήφισαν αυτό το, αυτή τη γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφαριών ε, πράγμα το οποίο επιβεβαιώνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να βοηθήσουν τις φτωχότερες περιοχές αλλά ακόμη και τις πιο πλούσιες και θεωρούμε ότι η πολιτική αυτή λειτουργεί σωστά και αυτό πρέπει να αλεχθεί σαφώς και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προς όλες τις κατευθύνσεις δηλαδή να μην υποβαθμιστεί η ε, πολιτική συνοχής για τις περιοχές οι οποίες ε, προχωρούν σωστά η Κωνσταντσα ε, τώρα παρακαλώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συγητή για το εξαιρετικό έγγραφο που κατήρτισε και δεν θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ήδη ο σκιώδης συγητής μας και τα οποία στηρίζω πλήρως. Έχω μόνο μία ερώτηση αρχή την οποία είχα θέσει και εχθές στους συντονιστές. Ανησυχώ πάρα πολύ και αυτό ε, διαδικαστικά πρέπει να διευκρινιστεί. Όταν διαπραγματευόμαστε τις προοπτικές, ε, διαπραγματευόμαστε θέματα που δεν έχουν ακόμη αποφασιστεί για την πολιτική συνοχή και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εισηγητής να έχει υιοθετήσει τις θέσεις μας αλλά θα αποφασίσει στο Συμβούλιο κατά τις διαπραγματεύσεις εάν πρόκειται να αποδεχθούμε μια θεματική ενότητα ή όχι. Αυτή η εντολή θα έπρεπε να διευκρινιστεί διότι νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν ε, περιλαμβανόταν στην έκθεση Γαρίγκα όπου η διατύπωση ήταν πολύ πιο γενική. Εκεί μιλάμε περισσότερο για τα συνολικά ποσά και ότι πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της ε, πολιτικής συνοχής. Αλλά πρώτη φορά ακούω ότι μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια ήδη στην MFF θα προσπαθήσουμε στο πολιετές χρηματοδοτικό πλαίσιο θα προσπαθήσουμε ε, να τα αποφασίσουμε όλα. Θα πρέπει εκεί να ασχοληθούμε και να διατηρήσουμε τις θέσεις μας στην διαδικασία συναποφάσεως διότι πολύ σωστά είπε ο εισηγητής ότι δεν πρέπει στο τέλος απλώς να μπορούμε να συνενέσουμε ή να αρνηθούμε θα πρέπει να μπορούμε να διαπραγματευτούμε. Ε, και δεν σημαίνει ότι δεν έχω ε, εμπιστοσύνη στον κύριο Κόβατσεφ ότι θα προασπιστεί τα συμφέροντα της, Επιτροπή, της Περιφερειακής Επιτροπής, αλλά θα πρέπει πάντοτε να σκέφτεται όταν διαπραγματεύεται ποιες είναι οι επιπτώσεις. Και γι' αυτό θα ήθελα ο εισηγητής για μια ακόμη φορά να ε, ελέγξει ακριβώς ποια είναι η εντολή και εάν δεν είναι σαφής πώς μπορούμε να ε, την διευκρινίσουμε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ τώρα να ε, στηρίξω τα σχόλια της Κωνσταντσα διότι πρέπει να δούμε εάν ε, η εντολή της Επιτροπής Προπολογισμού ήταν ακριβώς αυτή η οποία έπρεπε ε, διαφορετικά. Ναι μεν έπρεπε να αιτιολογήσει τους αριθμούς αναφέροντας τις πολιτικές αλλά όλοι έχουμε συμβάλει. Όχι μόνο η στην ψηφοφορία αλλά και στη συζήτηση. Πρέπει όμως να διευκρινιστεί πολύ σωστά ε, το ελέγχθη. Και στην Επιτροπή Προϋπολογισμού, εάν θέλουμε ε, να επηρεάσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ιουνίου ή Ιουλίου, διότι τότε θα υποβληθεί στο, ε, στη διάσκεψη κορυφής, θα πρέπει να έχουμε ψηφίσει εντός δύο μηνών για να είμαστε έτοιμοι για την Ολομέλεια. Δηλαδή πρέπει να δούμε τι θα γίνει με το ρυθμιστικό είναι ορισμένες πτυχές της εντολής που πρέπει να διευκρινιστούν. Δεν νομίζω ότι σήμερα ήδη έχουμε τις απαντήσεις και δίνω το λόγο τώρα στον Τόμας Ντόιτς. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή για το έγγραφο εργασία το οποίο μας εισηγήθηκε. Μας πάει και μας παρουσίασε. Πάρα πολύ α, θετικές αυτές οι νομοθετικές πρωτοβουλίες. Εγώ έχω δύο την να προσθέσω. να σας εξηγήσω ότι πρώτα πρώτα έχω πιστεί ότι οι ανταλλαγές απόψεων στην Επιτροπή μας τους τελευταίους μήνες μου δίνουν την εντύπωση ότι έχει χωριστεί στα δύο η Επιτροπή. Έχει χωριστεί στα δύο και παρουσιάζει το κάθε τμήμα της Επιτροπής διαφορετικά πράγματα, τελείως διαφορετικά. Ας πούμε οι μισοί παρουσιάζουν κάποιους στρατηγικούς στόχους, κατεβάζουν κάποιες προτάσεις. Να βοηθήσουν τον Επιτροποχάν. Και έρχεται ο, ο Επίτροπος και μας εξηγεί τους στρατηγικούς στόχους. Τους ε, στόχους για τους οποίους εμείς πάντοτε συμφωνούμε και υποστηρίζουμε. Όμως υπάρχει και άλλο ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο αγνοεί αυτούς τους στρατηγικούς στόχους. Έχουν άλλες συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις ας πούμε για το πολιτές ε, πλαίσιο. Είναι σαν ε, να μην συνδέεται το ένα τμήμα με το άλλο, δηλαδή σαν να μην συνδέονται καθόλου οι προτάσεις με την στρατηγική. Όπως τα έχουμε ακούσει εδώ, σε σχέση με την πολιτική της συνοχής. Υπάρχει τώρα ένα άλλο θέμα. Επηρεάζει η Περιφερειακή Επιτροπή την πολιτική της συνοχής και της αποφάσεις που λαμβάνεται. Η ουσία είναι ότι εάν έτσι συνεχιστούν τα πράγματα όπως πάνε, τότε οι διαπραγματευτές για τον προϋπολογισμό πρόκειται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση βέβαια και θα πρέπει εμείς να αποφασίσουμε για κάποια βασικά σημεία της πολιτικής συνοχής. Αλλιώς δεν θα επηρεάσουμε καθόλου το γίγνεσθε όσον αφορά τον καινούργιο προπολογισμό και την ε, περιφερειακή πολιτική. Όλα αυτά σα τα λέω γιατί θα έπρεπε στόχοι και λύσεις να συνδέονται. Σύμφωνοι. Χρειάζονται στρατηγικές ή γενικές, αλλά συγκεκριμένες λύσεις επίσης χρειάζονται. Θα πρέπει να λαμβάνετε περισσότερη υπόψη η γενικες αλλα συγκεκριμένε λυσεις επισης χρειαζονται θα πρεπει να βαλετε περισσοτερη υποψη η γνωμη τη Επιτροπή μα. Τώρα κάτι άλλο που είπε ο κ. Κόβατσεφ. Εγώ θεωρώ ότι έχει δίκιο και για τα τέσσερα σημεία που ανέφερε στην ε, εισαγωγή που μα έκανε. όσον αφορά την βοήθεια προς τα διάφορα κρατημέλη, όσον αφορά την συνοχή. Πώς δηλαδή θα μεγιστοποιηθεί αυτή η στήριξη σε σχέση με αυτό το 2,5% του ΑΕΠ που είναι απαράδεκτο. Πρόκειται για κάποια λύση, πρόταση που είναι ασυμβίβαστη σε σχέση με τους στρατηγικούς στόχους που έχει τάξει η ίδια η Επιτροπή. Σύμφωνα με τις ανησυχίες του εισηγητήριου στον αφορά την θεματική συγκέντρωση, είναι πολύ σημαντικά όσο μας είπε σε σχέση με την ευελιξία. Εδώ πέφτουμε σε αντιφάσεις. Ο κ. Άλμπρεχτ επίσης πολλές φορές μας έχει εξηγήσει ότι έχουμε διάφορες ε, διευκολύνσεις, διάφορες υποδομές όπως και αυτή που αφορά την διασύνδεση της Ευρώπης ε, έχουμε εδώ να οδηγούν σε κάποια σειρά λύσεων ανάλογα με την κατηγορία αλλά θα πρέπει οι προτινόμενες λύσεις να είναι ξεκάθαρες και άρα όταν δεν υπάρχει σαφήνεια δυσκολεύονται τα πράγματα. Άρα, θα πρέπει στατικοί και στατικοί στόχοι να συμφωνούν τα μεν με τα δε. Και να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες λύσεις. Πάρα πολύ στο είπε ο Γιώργος Κόβατσεφ. Πρόεδρος, εδώ θα κλείσουν κατά τον αγροτών συναδελφοί. Γιατί έχουν ζητήσει το λόγο έξι. Έξι συναδελφοί. Οπότε εδώ θα κλείσει η λίστα. Άρα πρέπει να ψηφορίες και άρα θα έχουμε δύο λεπτά να ομιλείτε. Δύο ο καθένας. Συγγνώμη, αλλά χτες μίλησαν... Ε, 20 δεν μιλήσανε, γιατί αυτοί που μίλησαν οι πρώτοι μίλησαν πάρα πολύ. Λάμπερ. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ πράγματι. Πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να είμαστε και τόσο αρνητικοί, διότι ε, βλέπουμε ότι έχουμε τουλάχιστον μία πρόταση από την Κομισιόν, η οποία αν δεν είχε υποβληθεί θα τις είχαμε ασκήσει σκληρές κριτικές. Έχουμε λοιπόν μία βάση, έχουμε μια αφετηρία με καλές προτάσεις. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά τα έγγραφα εργασίας. Εχθές μιλήσαμε πάρα πολλές φορές ε, για την ευελιξία, για τη θεματολογική συγκέντρωση. Ε, συζητήσαμε τις αρχές. Πρέπει να δούμε όμως ποια είναι τα διάφορα στοιχεία που θα μπορούσαν να απαντηθούν από την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εμείς θέσαμε πολλές ερωτήσεις. Τι ίδιες ερωτήσεις όμως πρέπει να τις θέσει και η Επιτροπή Προϋπολογισμών. Τώρα υπάρχει το πρόβλημα του κάπινγκ των οροφών μεταξύ των κρατών μελών, γιατί υπάρχει τέτοια μεγάλη διαφορά μεταξύ 2014-2020. Αυτό είναι ένα τυπικό παράδειγμα και θα πρέπει να επιμείνουμε για να μας δοθούν οι συγκεκριμένες απαντήσεις. Ας επιμείνουμε για μια ακόμη φορά ότι αν δεν έχουμε απάντηση δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε τόσα επίπεδα. Εμείς είμαστε εδώ στο Κοινοβούλιο, έχουμε συναδέλφους ε, σε διάφορες πολιτικές ομάδες οι οποίοι μπορεί να είναι συνομιλητές μας. Είπα ότι χθε ότι υπάρχουν διάφορες διαπραγματευτικές φάσεις. Θα πρέπει να συζητήσουμε με τον Λαμασούρ και με άλλους διότι αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εμείς ε, πρέπει να επενδύσουμε και στη διαδικασία. Ξέρετε ότι εδώ η γνωμοδότηση αποτελεί μόνο ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Ε, συζήτησα και με την Κωνσταντσα, πρέπει να συνεργαστούμε και με άλλους οι οποίοι πολλές φορές απουσιάζουν. Ας αναλάβουμε τις ευθύνες μας και ας συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι ε, πολύ σύντομος, αλλά δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε τη αρμοδιότητες της Επιτροπής Προπολογισμού χωρίς να εξετάσουμε τα θέματα της συνοχής και πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια να υπάρχει γενικά ένας μεγαλύτερος προϋπολογισμός. Δεν είναι μόνο θέμα συνοχής, αλλά χρειαζόμαστε γενικά ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Καταρχήν λοιπόν είναι το ποσό του προϋπολογισμού. Δεύτερον, οι στόχοι της πολιτικής συνοχής στον προπολογισμό. Είτε συμφωνούμε είτε όχι πρέπει να ενισχύσουμε τη θέση της συνοχής ε, στον προπολογισμό και όχι μόνο τη χρηματοδότηση. Τρίτον, υπάρχει ένα σημείο αμφιλεγόμενο σε αυτό το έγγραφο στο οποίο δεν θα συμφωνήσουν όλοι. Διότι η πρόταση να καθορίσουμε το 2,5% του ΑΕΠ σημαίνει να αυξηθεί, να μην υπάρξει πλαφόν, να υπάρχει διαφορετικό πλαφόν για διάφορες χώρες. Είναι διαφορετικές οι απαντήσεις. Δεύτερον, ο εισηγητής λέει ότι το 5% από το απόθεμα ε, για απόδοση performance reserve ε, ε, δεν είναι σωστό για το 5% αυτό. Συμφωνούμε ή όχι. Τρίτον, ο εισηγητής λέγει ότι έχουμε ένα μέσο να εξασφαλίσουμε τις επενδύσεις μας. 20% για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Δεν συμφωνούμε όμως όλοι με αυτά και ε, θα πρέπει καταρχήν ε, να γνωμοδοτήσουμε επί του προπολογισμού να πούμε ότι βασικά θέλουμε να υπάρξει μεγαλύτερος προϋπολογισμός να αυξηθεί ο προϋπολογισμός στο θέμα της συνοχής και να μην επισέλθουμε σε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η, σήμερα το πρωί ε, είναι, έχουμε μία συζήτηση για το, Ευρωπα... για το Ηνωμένο Βασίλειο πράγμα όμως ε, είναι σαν να λέμε ότι είναι όλοι αντιβρετανοί ενώ δεν είναι όλοι στη Βρετανία αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν αυτό που ήθελα να πω είναι ένα-δύο πράγματα σχετικά ε, με τους τελευταίους τελευταίους προϋπολογισμούς διότι στους, τα δύο τελευταία χρόνια θελήσαμε ε, ε, να εξασφαλίσουμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα συμμετέχουμε στη διαπραγμάτευση του πολιετού δημοσιονομικού πλαισίου από την αρχή και όχι μόνο στο τέλος. Βλέπουμε όμως ότι τώρα όποτε συζητάμε ε, για το πολιετές πλαίσιο, το MFF, υπάρχει ένα δισταγμός και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι προτού συζητηθεί σε επίπεδο του Συμβουλίου διότι ε, δεν μπορούμε ε, να ε, συζητάμε έτσι για όλο τον προϋπολογισμό και για τον προϋπολογισμό του μέλλοντος διότι εδώ ο βασικός παράγων είναι τα κράτη-μέλη εκ των οποίων ορισμένα θα ζητήσουν είτε να παγώσουν προϋπολογισμός είτε να μειωθεί. Έχω δύο ορισμένε προτάσεις κρατών μελών για ε, την πολιτική συνοχή και ζητούν ε, για το 2013-2014 να περικοπεί, όχι απλώς να παγώσει ο προπολογισμό. Οπότε ε, όπως έχω πει και προηγουμένως πρέπει να δούμε πού θα, ε, ε, πώς θα διανεμηθούν τα ποσά όπου χρειάζεται ευελιξία αλλά αναφερέστε 5% για τις πόλεις, 5% για το απόθεμα, 5% για τις περιφέρειες μειώνεται η διαπραγματευτική μας ευελιξία και πρέπει όπως είπαμε στην Επιτροπή Προπολογισμού να υπάρχει ε, ε, ευελιξία και θέλουμε ε, νομίζω να συνεργαστούμε επ' αυτού με την Επιτροπή Προπολογισμού που είναι ο σύμμαχός μας κατά τρόπον ώστε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε συμμαχίες στα διάφορα θέματα που μας απασχολούν. Θα πρέπει να έχουμε συμμαχίες και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί πολλά από τα θέματα θα προκύψουν όταν θα συζητήσουμε ορισμένα από αυτά τα θέματα ιδίως με συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Η Κορνέλια Ένς τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, ο οποίος πολύ σαφώς είπε περί τίνος πρόκειτο. Συμφωνώ σε πολλά θέματα μαζί του και ίσως θα πρέπει να δούμε ε, και να αναπτύξουμε ανά περιοχή ε, τι συνεπάγεται και πόσο αντιπαραγωγικό είναι το κάθε μέτρο. Λοιπόν, ε, γι' αυτό προτού συνενέσουμε ή αρνηθούμε θα πρέπει να υπάρχει υπάρξει μία ενιαία συζήτηση με, με την Επιτροπή Προϋπολογισμού όπου θα συζητήσουμε από κοινού τα κρίσιμα σημεία και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ ε, διότι έχουν μία διαφορετική οπτική γωνία αυτοί που κοιτάζουν γενικά και σφαιρικά το θέμα από αυτούς που το κοιτάζουν πιο ειδικά. Και άρα αυτή η συζήτηση θα ήταν επικοδομητική. Επιπλέον αναφέρομαι στα νέα ε, ε, ε, οικονομικά μέσα ε, και έχω μία άποψη από αυτού, δηλαδή είμαστε υπέρ των ταμείων που θα βαίνουν για ανακαίνιση αλλά πρέπει να δούμε πού, πρέπει να συζητήσουμε ακριβώς σε τι χώρους θα δημιουργηθούν και πού όντως μπορούν να συμβάλλουν και να ανακαινήσουν ε, αυτά τα νέα ανακαινιστικά ταμεία. Όσον αφορά το μέλλον των πόρων της ε, συνοχής αντιλαμβάνομαι ότι κινδυνεύει ε, διότι εάν από τη μία πλευρά αφαιρέσουμε το πρόγραμμα Connecting Europe βλέπουμε ότι μειώνονται οι χώρες και οι πόροι που θα συμμετέχουν στο Σταμείο Συνοχής. Πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε εν ώψη των προκλήσεων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε επαρκούν οι πόροι μας, διότι σκεφτόμαστε το θέμα τη φτώχεια και άλλα. Τέλο για τις περιφέρειες που είναι σε μεταβατική φάση. Υπάρχει ένας αριθμός σχετικά με το πώ θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι ε, περιοχές σε μεταβατική κατάσταση. Δεν ε, έχω γνώμη εδώ εάν πρέπει να αυξηθεί το ποσό αυτό ή να μειωθεί. Πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά νομίζω ότι έχουμε επαρκή χρόνο για να γίνει αυτό. Thank you. Jens Nielsen, please. Tack så mycket, herr ordförande. If it's okay, I can speak Swedish? Yes, of course. Yeah? Herr ordförande. Det är första gången jag tar till orda som ny medlem. Jag ska vara väldigt kort. Det är naturligtvis så att om budgetförhandlingarna Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να μιλήσει σουηδικά. Ο... Δεν, δεν υπάρχει πιβό από τα σουηδικά. Ωραία, θα μιλήσω αγγλικά. Μιλήστε ελληνικά. Μπορείτε να μιλήσετε και ελληνικά, άμα θέλετε. <clears throat> Όχι, όχι, θα προσπαθήσω να μιλήσω αγγλικά. Λοιπόν, Εάν πρόκειται να καταρρεύσει η διαπραγμάτευση για τον προπολογισμό, θα πρέπει ίσως να εξετάσουμε διαφορετικά τον κανονισμό και εκεί η Κωνσταντς έχει δίκιο. Γιατί ε, στο μέλλον θα μιλήσω πολύ για τη Βόρεια Φιλανδία και τη Βόρεια Σουηδία, όχι όμως τώρα. Τώρα αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο εισηγητής και η κυρία Φλόρα από την Επιτροπή Περιφερειών ε, ε, είναι σαν μια ωραία μουσική που ακούω διότι πρέπει να προασπίσουμε την, την ε, πολιτική συνοχής και πρέπει να πω ότι ένα από τα κράτη που θέλει να περιορίσει τον προπολογισμό είναι η Σουηδία και οι περιφέρειες στη Σουηδία στηρίζουν την Επιτροπή Περιφερειών και όχι τη Σουηδική Κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Γιένς, αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι εσύ θα πρέπει να αναλάβεις να αλλάξεις τη γνώμη της κυβέρνησή σου. Και τώρα ο Σον Κέλλη, τελευταίος ομιλητής. Ε, και εγώ θα μιλήσω αγγλικά και όχι την γλώσσα μου. Ε, και θέλω να κάνω γενικά σχόλια, διότι η Επιτροπή έχει ε, αναφέρει ότι η χρηματοδότηση πρέπει να ισχύσει παντού αλλά θα ήθελα να ρωτήσω εάν οι ε, πολίτες το γνωρίζουν και αν δεν το γνωρίζουν μήπως θα έπρεπε να το γνωρίζουν διότι εμείς δεν ε, έχουμε ε, την, τα ακούσματα από τους πολίτες για το πώς πρέπει να χρηματοδοτηθεί η Ευρώπη. Εφόσον λοιπόν είναι, είναι δικά τους τα χρήματα αυτοί πρέπει να υποφελούνται και ε, βλέπουμε ότι ε, δεν υπάρχουν ποτέ αμφισβητήσεις για πολύ αρνητικά θέματα. Ε, πολλές φορές, αν προσπαθήσω να αναστρέψω κάποια εξέλιξη αρνητική και πάω στον υπεύθυνο, μου λέει «Άστο, αγνόησέ το». Δεν είναι σωστό όμως αυτό, διότι για να προετύχουμε χρειαζόμαστε και δημόσιες σχέσεις και θα πρέπει στο μέλλον να αποδείξουμε ότι έγινε μία προσπάθεια να στηρίξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την χρηματοδότησή της και εν ονόματι των κρατών μελών και εν ονόματι των τελικών αποδεκτών. Ευχαριστώ. Προτού ζητήσω λοιπόν από τον Άντριο να σχολιάσω, θα ήθελα να σας πω τι κατάλαβα, που καταλήγω σχετικά με τα σχόλιά σας. Θέλουμε να εντοπίσουμε τα σημεία τα οποία θα έπρεπε ε, σαφώς να αναφέρονται στη θέση του Κοινοβουλίου και ε, πιστεύω ότι η εργασία σας για τις επόμενες εβδομάδες ε, θα πρέπει ε, να αποδείξει τι άλλο χρειάζεται. Τώρα έχετε το λόγο κύριε Κόβατσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι το εναρκτήριο έγγραφο δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο σχετικά με τον καθορισμό του επίπεδου για το 5% δεν υπάρχει μαθηματικός τύπος. Δεν ξέρουμε, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρει γιατί καθόρισε σαν όριο το 5%. Βεβαίως όσον αφορά το απόθεμα αποδοτικότητος, performance reserve, δεν ξέρω πώς καταλήξαμε σε αυτό και δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να υποφέρει μία περιοχή, γιατί η άλλη τα καταφέρνει καλύτερα για πολιτικούς λόγους ή άλλους. Μετά, πολύ καλό και πολύ σημαντικό θέμα κυρία Κέλ. Ε, είναι ποιος έρχεται πρώτος, ε, το αυγό ή το κοτόπουλο. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να διευκρινιστεί στην Επιτροπή. Ε, όσον αφορά τους κανονισμούς και το διοικητικό πακέτο, πρέπει να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες. Συμφωνώ μαζί σας, πρέπει να διευκρινίσουμε ε, την εντολή με την Επιτροπή ε, Προϋπολογισμού σχετικά με το πολιετές οικονομικό πλαίσιο και πού μπορούν να προβούν σε ρυθμίσεις και πού μπορούν να αποφασίζουν ε, την πολιτική συνοχή από πλευράς ε, προϋπολογισμού. Εδώ λοιπόν κυρία Πρόεδρε θα ήθελα τη στήριξή σας. Ίσως ε, θα έπρεπε όπως ελέγχθη από συναδέλφους να κάνουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ επιπλέον για όλες τις επενδύσεις θα ήθελα να συνεχίσουμε τώρα στα θέματα τα οποία έχουμε εντοπίσει, να διαγράψουμε κατευθύνσεις για μεγαλύτερα ποσοστά, μαθηματικές, μαθηματικές συγκεντρώσεις, τέλος πάντων να καταρτήσουμε μία κοινή θέση της Επιτροπής και να μπορέσουμε να τη μεταδώσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμού. Άρα δεν χρειάζεται άλλη απόφαση επί του θέματος αυτού, απλώς θα συνεχίσουμε την εργασία με, προς την κατεύθυνση που διαγράφηκε στη συζήτηση και τώρα θα ήθελα να ψηφίσουμε καταρχήν να δείτε αν τα μηχανήματά σας δουλεύουν σωστά. Ah,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 Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παρακαλώ βάλτε ε, τα ακουστικά σας για να ελέγξουμε το σύστημα. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι ο Μάρκους να καθίσει. Λοιπόν, ξεκινάει η ψηφοφορία για να ελέγξουμε το σύστημα. Οπότε σε δύο λεπτά θα σταματήσουμε την ψηφοφορία. Όλοι έλεγξαν τα μηχανήματά τους. Νομίζω ότι πήγαμε καλά, οπότε σταματάει η ψηφοφορία, η δοκιμαστική τώρα. Και προχωράμε στην ε, πρώτη ψηφοφορία για το μέλλον των περιφερειακών αεροδρομίων της κυρίας Σούτζας και ξεκινάμε με την πρώτη συμβιβαστική. Ε, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 9. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερη συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 16 υπάρχει μία προφορική τροπολογία ε, είναι κανείς αντίθετο στην ε, ε, προφορική τροπολογία όχι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 35 We have to check. πρέπει να ελέγξουμε την ε, τροπολογία 35 ξεκινάει η ψηφοφορία Closed. πέρας της και απορρίπτεται 26-19. Πάμε τώρα στη συμβαστική υπερθυμών 6. Ποιοι είναι υπέρ. Αλλά. Το μικρόφωνο σου, Αλένα, λες τον κύριο Καντέκ. Για τον συμβιβασμό 35. Έχουμε κάνει λάθος και ο Μπρίς και εγώ κάναμε και οι δυο λάθος, ήμασταν υπέρ. Δεν αλλάζει τίποτα, αλλά να το ξέρετε έτσι γενικώ για, την ιστορία να πούνε σε 20-25 χρόνια ορίστε ψήφισαν υπέρ. Συμβιβασμό 6 αγαπητοί συνάδελφοι, Ποιο είναι υπέρ κατά. Αποχές, εγκρίνεται και πάμε τώρα στην τροπολογία 43. Ποιο είναι υπέρ, ποιο είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα για την ε, τελική συνολική ψηφοφορία ηλεκτρονικά και ψηφίζουμε. Πέρας. 41 1 3. Congratulations. ένα, αποχές. Συγχαρητήρια. Και τώρα θα πάμε στη δεύτερη ψηφοφορία. Αφορά τη διαχείριση της ποιότητας των στατιστικών. Λουκατσίευσκα είναι η συγγήτρια. Εδώ έχουμε ε, μια τροπολογία του κυρίου Μπεσέ. Και ψηφίζουμε όπως τροποποιήθηκε προφορικά. Υπέρ, κατά. Οπότε συγκρίνεται και υπάρχει μια προφορική ε, για την παράγραφο 4. Υπέρ, κατά. Ψηφίζουμε. Αποχές, εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Λαμπέρ. Πώς θα ψηφίσουμε. 44-1 εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Πάρα πολύ γρήγορα τα πήγαμε και πάμε στο επόμενο. Είναι έκθεση Μπέρντερ. Δύο ποικιλότητα για το 2020. Η συγγήτρια έχει στο λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μισό λεπτό. Ελπίζω δεν είπα κάτι και πείραξε τον κόσμο και φύγαν όλοι. Έχουμε επομένω ε, αυτή την ανακοίνωση για τη βιοπικιλότητα 2020 που το όνομα 2011 πρώτα πρώτα εξεδόθηκε. Πρόκειται για μέρο τη στρατηγική για το 2020 για το θέμα αποτελεσματικού, αποτελεσματικότητα των ε, πόρων και έχει πάρα πολλά ενδιαφέροντα εδώ όσον αφορά την καταπολέμηση τη αλλαγή του κλίματος, ε, γιατί εδώ έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τις επιδόσεις μας και έχουμε, έχω μια γνωμοδότηση στην Τροπή Περιβάλλοντος που τα έχετε, έχετε λάβει το κείμενό μου οπότε θα θέλω και εγώ τώρα να σας πω τις σκέψεις μου σχετικά πρώτα πρώτα έχουμε την παραγραφή υπαριθμών 1 που λέει για την απόλυτη ποικιλότητα τι απειλέ, ε, από τα χώρα κατακριτικά είδη, υπερκατανάλωση φυσικών πόρων, ότι όλα αυτά το τα λέμε η, λέμε η σιωπηλή κρίση. Γιατί όλα αυτά θα έχουν πάρα πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής όλων μας. Οπότε κατεπηγόντως χρειάζεται να ληφθεί δράση σε κάθε επίπεδο. Δεύτερον, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να ε, ε, λάβετε υπόψη το ότι οι πόλεις. Είναι απειλή αλλά και καταφύγιο. Άρα θα πρέπει να αναγνωριστεί η σχετική πολιτική. Η χωροταξία, ο προγραμματισμός σε σχέση με τις πόλεις και αυτά τα λέω στην παράγραφο 2 της εκθεσιός μου. Επίσης, θεώρησα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε σε αυτή τη συγκυρία της οικονομικής αβεβαιότητας ότι πολλές φορές δεν θεωρείται προτεραιότητα το περιβάλλον, ότι θα πρέπει να προσέξουμε την πράσινη οικονομία διότι βοηθά για να έχουμε κατάρτιση ε, ε, και τις δεξιότητες και όπως όλα αυτά τα είπε το πόσο οφείλεται την οικονομία, η πράσινη οικονομία ο Δανός υπουργό, οπότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη πόσο σημαντική είναι η βιοπικιλότητα και θα πρέπει οι τοπικές περιφερειακές αρχές να βοηθήσουν ε, και να εμπλακούν στη διαδικασία λήψη αποφάσεων, γιατί πολύ συχνά ρίχνουμε την ε, προσοχή μα στην ανάπτυξη και ξεχνούμε την παραδοσιακή γνώση που, όπου θα πρέπει να την εγκαλιάσουμε για αυτήν και τέλο τα, τα, τα κέρδη από την προστασία τη βιοπικιλότητα ε, εμπλέκουν μη κυβερνητικέ οργανώσει, θέλοντέ, θα πρέπει να του ενθαρρύνουν να συνεχίσουν να αποτελούν τμήμα για την, την, την, την της πολιτικής μας, όπως θα πρέπει την Μαρίνα Πέντζεβα να την ευχαριστήσω ε, και την Ταϊάννα Χάς, την υπάλληλο της Επιτροπής μας, γιατί με βοήθησαν πάρα πολύ και επίσης περιμένω να ακούσω τις απόψεις συνάδελφοι για το σημαντικό τούτο θέμα. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ε, εσείς εκπροσωπείτε τον Μάρκος. Ο συνάδελφος Κούρια, κυρία Πρόεδρε, δεν είναι πια μέλος αυτής της Επιτροπής. Και προσεκλήθην εγώ να τον αντικαταστήσω για την έκθεση ως σκιώδης εισηγητής. Εγώ ευχαριστώ τη συνάδελφο για την γνωμοδότηση. Εγώ πιστεύω ότι αυτό το έγγραφο είναι πάρα πολύ σημαντικό για τις, για τις εργασίες της Επιτροπής μας. Το ουσιαστικό σημείο των εργασιών μας είναι η τεκμηρίωση της δαπάνης βάσει των κριτηρίων της, ε, ε, του δημοσιονομικού πλαισίου της Κομισιόν και το περιβάλλον και όλα τα παρεμφερή θέματα ε, εντάσσονται σε αυτήν την οπτική και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Επιτροπή επί της ουσίας να λάβει υπόψη τις υποδείξεις που εμείς θα υποβάλουμε. Κυρίως όσον αφορά ε, στο περιβάλλον και τον καθορισμό προτεραιοτήτων ε, και εμπλοκών που έχουμε στην επικράτεια. Και εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να προσέξουμε όλες τις δράσεις που εντάσσονται στην αστική ατζέντα, στην ατζέντα για τις πόλεις. Και μέσα σε αυτήν θα πρέπει να υπάρχει και μία ένδειξη για το ποια μέτρα υπερισχύουν, δηλαδή τα μέτρα εκείνα που καθιστούν συμβατή την ανάπτυξη με την περιβαλλοντική ισορροπία, δηλαδή με οικοαϊφόρους στόχους. Εγώ θέλω να συγχαρώ τη συνάδελφο για, τις εργασίες, για τη δουλειά της. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτή την έκθεση στη συνέχεια, ούτω ώστε η πρόταση της Περιφερειακής Επιτροπής προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος να είναι πιο χρήσιμη και πιο πλήρης. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Ο Λέινιτσακ, όχι, δεν θέλεις τον λόγο, είσαι σκιώδης ηγητής. Συγγνώμη, ε, είχα, ε, ήμουν αφηρημένος, έκανα άλλα πράγματα. Εγώ ήθελα να πω το εξής για αυτά τα οποία συζητάμε. Δεν έχουμε σχόλια. Υποστηρίζουμε πλήρως την πρόταση η οποία κατατέθηκε και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος για Κύριε Πρόεδρε, ε, θα θέλαμε και εμείς να ευχαριστήσουμε την κυρία Μπέρντερ για τη γνωμοδότηση που είναι πολύ καλή, έχει θετικά στοιχεία. Θα ήθελα να αναφέρω όσον αφορά την ε, προηγούμενη στρατηγική για την ε, βιοπικιλότητα, η οποία απέτυχε εντελώς στην εφαρμογή. Θα πρέπει να προσθέσω ότι εμείς ως πράσινοι χαιρετίζουμε τις προϋποθέσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο πριν ξεκινήσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα κάποιοι συγκεκριμένοι μηχανισμοί πρέπει να εφαρμοστούν να τρέξουν ώστε να γίνει πιο ορθολογικός έλεγχος. Επίσης, οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να γίνουν εθνική νομοθεσία. Οι περιβαλλοντικές δοκιμές συμβατότητας είναι αναγκαίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης στρατηγικής πρέπει να τεθούν κριτήρια αξιολόγηση Δύο λόγια για την Ελλάδα όπου η Επιτροπή φαίνεται να χάνει τη μάχη για την προστασία της βιοποικιλότητας, Καθώς οι νόμοι αλλάζουν, οι κανόνες δεν λαμβάνονται υπόψη, υπάρχει η διαδικασία του fast track. Εχθές είχα τη διάθεση να κάνω αυτή την ερώτηση και στον Επίτροπο τον κύριο Χάν, γιατί μίλησε για την προστασία ε, των περιοχών Natura, αλλά δεν έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για μέτρα. Όταν λοιπόν η Ελλάδα βουλιάζει στην κρίση και λόγω των σχεδιαζόμενων έργων βλέπουμε ότι υπάρχει αντίληψη ότι θα προωθηθούν οι δείκτες της οικονομίας αλλά χωρίς να παίρνετε υπόψη το περιβάλλον σημαίνει ότι θα έχουμε υψηλό περιβαλλοντικό κόστος. Τα κονδύλια δεν πρέπει να χορηγούνται με στόχο μόνο οικονομικό αλλά για την προστασία της βιοπικιλότητας. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τόνωση της οικονομίας χωρίς να παίρνουμε υπόψη και άλλους παράγοντες. Με αυτές τις παρατηρήσεις κλείνω επαναλαμβάνοντας ότι έχουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. λόγω του πρωτοπόρου έργου των πράσινων ο κόσμος κατάλαβε ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα και αυτό αποδείχθηκε σήμερα για το πώς ενδιαφέρονται όλες οι πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Τώρα, έχω δύο τι να, να σας αναφέρω. Αυτή η ανοιχτή ατζέντα είναι πάρα πολύ σημαντική για την βιοποικιλότητα θα πρέπει να καλυφθούν όλοι και όχι μόνο οι Πέτρος. Τώρα, σε σχέση με τα ανοιχτά σχολεία και τους μαθητές που θα πρέπει να διαπιστώνουν, να νιώθουν, να έχουν την εμπειρία της βιοποικιλότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα πρέπει λοιπόν και αυτό εγκαίρως να καλυφθεί. Κάτι άλλο το οποίο είπε η Κατερίνα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μας μίλησε για το ότι χρειάζεται να εμπλέξουμε ε, τις κοινότητες, τις ε, τοπικές αρχές, τους εθελοντές και έχει δίκιο γιατί από πολλέ πλευρές αυτοί είναι οι φυσικοί πρωταγωνιστές πάνω σε αυτό, πάνω στον αγώνα για τη βιοπικιλότητα στην κοινωνία. Άρα μέσω αυτών θα εμπλακεί και η κοινωνία είναι καλό αυτό και ο πλευρά τη πολιτική. Άρα, το κείμενο αυτό έχει σωστέ σκέψει και πάνω σε αυτέ αξίζει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Εμεί ευχαριστούμε. Δεν έχουν ζητήσει άλλο το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την γνωμοδότηση. Κατα... Είμαστε στη φάση 2 συν 20. Στο Ρίο είχαν υπογραφεί δύο πρωτόκολλα, ένα για, το, για την κλιματική αλλαγή και ένα για τη βιοπικιλότητα. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι προχώρησε ιδιαίτερα γρήγορα η συνειδητοποίηση των προβλημάτων στον τομέα της κλιματικής αλλαγής αλλά όχι της βιοποικιλότητας, που είναι εξίσου σοβαρή αν όχι περισσότερο διότι βρισκόμαστε στο, εξ, στο έκτο κύμα εξαφάνισης των ειδών. Πρέπει λοιπόν η Ένωση να στοχεύσει και στις υπερπεριφερειακές περιοχές διότι το μεγαλύτερο ποσοστό της βιοπικιλότητας βρίσκεται στις υπερπόντιες περιοχές. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή των συναδέλφων μου σχετικά με την εφαρμογή του Natura 2000 γιατί το Natura 2000 δεν εφαρμόζεται στις γαλλικές υπερπόντιες περιοχές και αυτό για διάφορους λόγους άγνωστους όμως και θολούς. Χρειάζομαι λοιπόν την υποστήριξη των συναδέλφων για να υποστηρίξω μία τροπολογία που θα καταθέσω ούτως ώστε να καλύψουμε αυτό το κενό. Νίκολσον. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα πρώτα απ' να συγχαρώ την εισηγήτρια. Να σας πω ότι συμφωνώ μαζί της τότε που μας είπε για αυτήν την σιωπηλή κρίση πάρα πολύ εύγλωτα διατυπώνει τα πράγματα έτσι. Πολύ σημαντική και αυτή η ατζέντα για τις πόλεις. Όντως τα παιδιά θα πρέπει να δουν τα υπέρ και τα κατά της βιοποικιλότητας και όχι μόνο να βλέπουν τα θέματα αυτοί που ζουν στην Ήπεθρο. Όντως θα πρέπει να προστατεύσουν το περιβάλλον. Είναι κορυφαία προτεραιότητα. Θα πρέπει επομένω να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Μη και κυβερνητικέ οργανώσει, εθελοντέ και αυτοί να εμπλακούν, όντω. Ε, πρέπει να του βοηθήσουμε. Είναι, έχουν ήδη που δεν χρειάζεται να του εμπλέξουμε. Όμω, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις τοπικές αρχές, μια που αυτή είναι πιο κοντά στο πρόβλημα. Αυτοί μπορούν να εντοπίσουν τις ανάγκες τους και άκουσα τα θέματα από ε, την κάθε χώρα και κάθε χώρα έχει διαφορετικά προβλήματα. Άλλα έχει η Ελλάδα, αλλά έχουμε εμείς τη χώρα μας. Γι' αυτό και χρειάζεται οι τοπικές αρχές να εμπλακούν. Επομένως, γι' αυτό σας λέω ότι πάρα πολύ καλά τα πήγε η συγγήτρια. Κύριε έχετε Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια για το κείμενο το οποίο πρότεινε σήμερα. Θα ήθελα όμως να της ε, αναφέρω μία τροπολογία και αυτό για μία θέση που ήδη έχει αποφασίσει το κοινοβούλιο μας με μεγάλη πλειοψηφία για την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Το Συμβούλιο θα ήθελε να περιορίσει ε, και οι Κομισιόν θα ήθελαν να περιορίσουν την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων ε, οργανισμών. Αν επαναλάβουμε εμείς αυτή την αρχή και μέσα στο κείμενο, τότε θα επαναλάβουμε την θέλησή μας, τη βούλησή μας που αποτελεί ε, εγγύηση για το μέλλον και των γενεών μας και για την εγγύηση της βιοπικιλότητας που είναι ο πλούτος μας. Καταλαβαίνω ότι ήσασταν ο τελευταίος, η Κατρίν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ όλους για τα όσα είπατε. Νομίζω ότι πάρα πολύ θετικά. Ε, πάρα πολύ ευχάριστο να ξέρω ότι οι συνάδελφοι με στηρίζουν. Τώρα, τα κριτήρια για τις δαπάνες είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα πρέπει να ντρεπόμαστε γιατί ε, απέτυχαν οι προηγούμενες ε, στρατηγικές. Γιατί είπαμε ότι έχουμε την ε, μία κρίση που μπορεί να κρύβει την άλλη. Δηλαδή δεν ωφελεί να ανθεί η οικονομία όταν έχουμε κρίση περιβαλλοντική απώλεια ποικιλότητα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν. Και θα πρέπει να δούμε πώς όλα αυτά θα μπορέσουμε να τα περάσουμε στις τοπικές αρχές, τοπικά δίκτυα, με τις μη κυβερνικές οργανώσεις, ε, δημοτικές αρχές. Εκείνοι είναι εκεί, εκείνοι θα εφαρμόσουν την πολιτική. Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι η πληθώρα των διαφορετικών κατηγοριών προστατευμένων περιοχών. Για να δούμε τώρα, περιμένω τις ε, τροπολογίες. Ε, εμείς ευχαριστούμε τον πρόεδρο και τώρα η απόφαση που πρέπει να λάβουμε είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και εγώ θα ήθελα επίσης να σας ε, προτείνω ε, Ε, το Φεβρουάριο τέλο πάντων. Πάμε τώρα στην έκθεση Deutsch όσον αφορά το τρίτο τμήμα. Το τρίτο τμήμα για τον προπολογισμό που αφορά την Επιτροπή. Τμήμα 3. Τόμας Deutsch, έχει το λόγο. Συνάδελφοι, επιτρέψτε μου να σας πω με συντομία τις παρατηρήσεις μου. Ε, τα βασικά τα έχετε λάβει στο φαγγελό σας και τι θα ήθελα πρώτα πρώτα να σας αναφέρω ότι είναι πάρα πολύ βασικό να λάβετε υπόψη ότι θα πρέπει να τοποθετηθούμε όσον αφορά την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προπολογισμό και θα πρέπει να προσέξουμε εδώ το τι θα γίνει με την πολιτική της συνοχής και τη διαχείρισή της. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ε, ενδιαφέρει πάρα πολύ την Επιτροπή μας. Ακούσατε προηγουμένως Τι έχει προηγηθεί τόσα χρόνια. Τις οικονομικές αβεβαιότητες. Ξέρουμε ότι τώρα σώβει μια κρίση. Υπάρχει και κρίση εμπιστοσύνης. χάσαμε την εμπιστοσύνη που είχαν οι Ευρωπαίοι στο πρόσωπό μας επομένως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε ακόμα περισσότερο ε, το πώς θα δαπανώνται τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Να γίνεται δηλαδή αυτό με προσοχή διαφάνεια, οπότε και για την απαλλαγή του 2010 ισχύουν όλα αυτά. Και σε σχέση με το 2009 3, από 3,3 πήγε σε 3,7 το ποσοστό σφάλματος. Ο κόσμος θεωρεί υπεύθυνη την πολιτική συνοχή. Θα πρέπει εμείς όμως κάτι να κάνουμε τόσο να αντικρούσουμε τα επιχειρήματα αυτά τα οποία αποτελούν κατηγορίε επικρίση για την πολιτική συνοχή. Σε αυτό κάνω και εγώ στο κείμενό μου και έχουμε δεδομένη και την έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Εκεί συζητάμε για την εκτέλεση του προπολογισμού στη σχετική περίοδο. Έχουμε την περίοδο προγραμματισμού 2007-2011 κατά την οποία περίοδο αυτή η χρήση του 2010 δηλαδή ήταν ε, η πρώτη περίπτωση, η πρώτη φορά κατά την οποία δόθηκαν τόσα πολλά χρήματα στην ε, πολιτική συνοχή. Βεβαίως και η πολιτική της συνοχής είναι η πολιτική η οποία επιδέχεται τα περισσότερα σφάλματα κατά την υλοποίησή της. Αυτό αναφέρει και η έκθεση του Ελληνικού Συνεδρίου. Άρα θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη. Γιατί σε σχέση με την περίοδο 2002-2006 το επίπεδο σφάλματος μειώθηκε και τη χρήση 2009 και τη χρήση 2010 είχαμε μικρότερο επίπεδο σφαλμάτων. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, αλλά βέβαια ε, δεν θα πρέπει να υπαραπαυτούμε γιατί συνεχίζει και υπάρχει αρκετά υψηλό επίπεδο ασφαλμάτων. Ε, Τα σχετικά σφάλματα συνήθως αφορούν προμήθειες, διαγωνισμούς, δημόσιες συμβάσεις. Και άρα θα πρέπει να προσέξουμε τους κανόνες επιλεξιμότητας, τους κανόνες που διέπουν αυτές ε, τις δημόσιες συμβάσεις. Και ο κόσμος επομένως συνεχίζει και ισχυρίζεται ότι χρειάζεται περαιτέρω απλούστευση των σχετικών διαδικασιών και αυτό το προσέξουμε σε σχέση με την φετινή απαλλαγή πάρα πολύ σημαντικό αυτό το μήνυμα να το στείλουμε ξεκάθαρα. Κάτι άλλο τώρα. Το οποίο αφορά το ελεγκτικό συνέδριο, την έκθεσή του. Περισσότερες ε, πράξεις πάσχουν. Υπάρχουν πολλά σφάλματα αυτές οι πράξεις και συναλλαγές δηλαδή που αφορούν τις εθνικές αρχές και έχουν ζητήσει τους όλα τα μέσα που χρειάζονται οι εθνικές αρχές ούτως ώστε να διορθώσουν την κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά την συνδιαχείριση, δεν ε, φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι φτάνει οι εθνικές αρχές που ακριβώς μπόρεσαν, δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα που διαθέσει την διευθυντική κατάσταση. Γιώργος Σταυρακάκη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότηση που μόλις τώρα μας παρουσίασε, το οποίο πιστεύω αποτελεί μια πολύ καλή βάση και πάνω σε αυτή τα δουλέψαμε. Για το οικονομικό έτος 2010 και πάλι η πολιτική συνοχή βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης, κύρια όσον αφορά το ποσοστό λάθους και το αντίκτυπο που έχει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι διαπιστώθηκε μια καλύτερη κατάσταση από εκείνη της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου 2000 2006. Ωστόσο, πρέπει να, είμαστε, να έχουμε μια σαφή εικόνα και να υπογραμμίζουμε τι συνιστά λάθος και τι όχι. Λάθος συνιστά μια συναλλαγή που δεν συνάδει στο σύνολό της με τους ισχύοντες κανονισμούς. Λάθος όμως από την άλλη πλευρά δεν σημαίνει ότι οι πόροι έχουν χαθεί ή έχουν σπαταληθεί ή ότι έχει διαπραχθεί απάτη. Επιπλέον, τα στοιχεία δείχνουν ότι τα δύο τρίτα των λαθών επικεντρώνονται σε τρία από τα 27 κράτη-μέλη και σε 7 από τα 455 προγράμματα. Τούτο σημαίνει ότι με στοχευμένη προσπάθεια από την Επιτροπή και, τα συγκεκριμένα, και από τα συγκεκριμένα κράτη, το ποσοστό λάθους θα μπορούσε να μειωθεί σημαντικά. Είμαι σίγουρος ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περίοδου στην πολιτική συνοχή θα πρέπει να υπάρξει ένας μεγαλύτερος βαθμός απλούστευσης και ελέγχων που συνδυάζουν αποτελεσματικότητα και κόστος το οποίο τελικά θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Thank you very much. Ramona Manescu, Ramona Manescu. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ντόιτς καταρχήν. Εγώ πιστεύω ότι για μια ακόμη φορά συνειδητοποιούμε ότι αυτά τα εφαρμοστικά λάθη έχουν τη ρίζα τους έχουν τη ρίζα τους το γεγονός ότι, ότι τα προγράμματα δεν ενσωμάτωσαν τις λύσεις που δώσαμε εμείς στο Κοινοβούλιο. Δηλαδή, αμάρτησαν λόγω υπερβολικής ε, ρυθμιστικότητας. Πρέπει λοιπόν να, να πλουστεύσουμε όλο αυτό το σύστημα οικονομικής μηχανικής. Το λέμε, το ξαναλέμε και δεν γίνεται ποτέ τίποτα και από αυτό γεννιούνται ένα σωρό προβλήματα. Κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την νομοθεσία. Αν καταφέρουμε να αλλάξουμε και το πνεύμα του δημοσίου, των δημοσίων υπηρεσιών, θα μπορέσουμε να λύσουμε πολλά προβλήματα γιατί πολλές φορές η βάση των λαθών βρίσκεται και στη διαφορετική ερμηνεία και αντιμετώπιση της κοινοτική νομοθεσίας από τη δημόσια διοίκηση στις χώρες. Δεν ζητήσει άλλη το... Α, όχι, όχι, όχι, συγγνώμη, Ναι, ναι, τη εγγραφή στον κατάλογο. Ο Φρανσουά, ευχαριστώ πρόεδρέ μου. Συμφωνώ απόλυτα με την ε, παρουσίαση του κυρίου Ντόιτς. Βέβαια θεωρώ ότι η γραπτή παρουσίαση ε, είναι αρκετά φτωχή, θα έπρεπε να είναι πιο, πιο δυναμική, θα έπρεπε ήδη να εκφράσετε και την ικανοποίησή σας για την μείωση του ποσοστού των λαθών, Πολλές φορές έχουμε ε, λάθη τα οποία δεν είναι λάθη επί της ουσίας, ότι τα περισσότερα λάθη θα μπορούσαν να λυθούν μέσα από τη διοικητική απλούστευση και μετά θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για το καλύτερο ποσοστό. Αυτό θα, νομίζω ότι θα έπρεπε να δοθεί από την Επιτροπή μας, να δοθεί ένας πιο, θετικό, πιο θετικός ε, τόνος. Ε, πολλές φορές η αυστηρότητα μπορεί να παγώνει τους ενδιαφερόμενους. <coughs> Και θα έπρεπε λοιπόν ο δημοσιονομικός έλεγχος να λάβει υπόψη όλη αυτή τη θετική δυναμική. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Τόμα, σε παρακαλώ μπορείς να σχολιάσεις. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, λέει ο κύριος Ντότς. Και θα ήθελα πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια, την προστηρίξή τους. Έχω τρία την να σας αναφέρω. Πρώτα-πρώτα ανέφερε ο Αντιπρόεδρος ε, Σταυρακάκης με τον οποίο και συμφωνώ πόσο σημαντικό είναι το ότι θα πρέπει να κάνουμε στο σημείο που ανέφερε μία τροπολογία. Έχουμε λοιπόν τρεις ε, κατηγορίες διαφορετικών ασφαλμάτων. Όταν υπάρχουν επομένω ε, επιπτώσεις οικονομικές, αυτό είναι μια διαφοροποίηση. Δηλαδή δεν συνιστά κάθε σφάλμα απάτη. Δεν το έχουν καταλάβει αυτό όλοι. Υπάρχει σύγχυση αρκετή. Όχι. Κάποια λάθη δεν συνιστούν απάτη. Γιατί υπάρχουν άλλωστε και κάποια σφάλματα που δεν έχουν κάνει οικονομικέ επιπτώσει. Κύριε Μανέσκο, πάντω μα ανέφερε ότι υπάρχουν κανόνε κοινοτικοί. Και μπορούμε να επιστρέψουμε αυτούς τους κανόνες για να προστέψουμε την κατάσταση. Όμως, ξέρετε, η επικουρικότητα κάνει τις εθνικές διατάξεις να κατησχύουν και δίνει επομένως τον μπαλάκι την πρωτοβουλία την προτεραιότητα στις εθνικές αρχές. Άρα θα πρέπει και εμείς να δούμε πώς μπορούμε την κατάσταση να την βελτιώσουμε. Συμφωνώ και σας ευχαριστούμε για τις πατρίες σας. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Η τροή προθεσμία είναι, όπως και στην προηγούμενη έκθεση, το μεσημέρι της Δευτέρας Φεβρουαρίου. Το μόνο σημείο τώρα της μέσης διατάξεως είναι και αυτό σχέδιο εκθέσεως της Βασιλίτσια Βιωρίτσα Ντάντσελα και αφορά το έκτο αλλά και έβδομο πρόγραμμα δράσης. Έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτό το πρόγραμμα συνεισέφερε πολύ σημαντικά στην περιβαλλοντική πολιτική της Ένωσης. Υπάρχει όμως πρόβλημα με την εφαρμογή. Και αυτό δηλαδή λόγω της ε, κρίσης ε, σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντική η προσπάθεια που γίνεται για να διευρύνουμε το Natura 2000 ε, και όλα όσα χρειάζονται για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Εγώ θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν θα έπρεπε να δράσουν από κοινού για να μπορέσουν να διαπιστώσουν όλους τους τομείς εκείνους όπου μπορεί να εφαρμοστεί καλύτερα η κοινοτική νομοθεσία και να μειώσουν τη διαφορά μεταξύ των στόχων του έκτου προγράμματος και του τελικού αποτελέσματος. Το έκτο πρόγραμμα ολοκληρώνεται στα μέσα του 2012. Πρέπει λοιπόν εμείς να φτιάξουμε ένα καινούριο πρόγραμμα που θα λαμβάνει υπόψη το τωρινό πλαίσιο αλλά και τις μελλοντικές εξελίξεις. Το έκτο πρόγραμμα δράσης θα μπορούσε να αποτελέσει μία νέα ευκαιρία για να λύσουμε τα προβλήματα και θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τον, την νομοθετική εστίαση με τη στρατηγική. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ε, και την πρόληψη είναι κάτι το πάρα πολύ θετικό η πρόληψη και αυτό θα μας οδηγήσει στο να καλύψουμε και την προβληματική των χώρων όπου το χώρο κατοικίας, δηλαδή θα πρέπει να διευρύνουμε όλες τις υπηρεσίες ε, για τον κόσμο, νοσοκομεία, σχολεία κλπ. Χρειαζόμαστε χώρο κατά συνέπεια. Οπότε οι αστικές περιοχές χρειάζονται νέους τρόπους ε, επέκτασης. Θα πρέπει επίσης να έχουμε όλους αυτούς τους νέους χώρους και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις όμορες υπαίθριες περιοχές. Θα χρειαστούν νομοθετικά μέτρα που να αλλάξουν τον προορισμό αυτών των ε, εδαφών. Τώρα περισσότερος πληθυσμός σημαίνει περισσότερη τροφή. Χρειάζεται μεγαλύτερη πίεση για το πώς θα χρησιμοποιείται η γεωργική γη. Χρειαζόμαστε λιγότερη ρήπανση από τα οχήματα όλων των τύπων και θα χρειαστούμε νέα πρωτότυπα που θα καταναλώνουν νέα καύσιμα. Με αυτά όμως τα νέα καύσιμα θα πρέπει να αλλάξουμε και τον προορισμό των χωραφιών θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις πολιτικές περιβάλλοντος και να τις συνδυάσουμε με τις πολιτικές υγείας και με άλλες πολιτικές. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε μία ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Όπως ανέφερα, πρέπει να σκεφτούμε και την πρόληψη και όχι μόνο το πώς θα διορθώσουμε όλα όσα, έχουν, ε, όσα χρειάζονται διόρθωμα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας όλες τις πλευρές. Αέρα, νερό, έδαφος. Θα πρέπει να βρούμε λύση για την ανακύκλωση των σκουπιδιών που θα είναι όλο ένα περισσότερα. Πρέπει να βρούμε ένα πρόγραμμα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Αν βρούμε μία σωστή διαχείριση θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε μέχρι και 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. και θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε πάνω από 4.000 εργασία, θέσεις εργασίας και αυτό είναι συμβατό με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Χρειάζεται λοιπόν να βελτιώσουμε τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών και αρχών και τοπικής αυτοδιοίκησης με τις κοινοτικές αρχές. Είναι πολύ σημαντικό, ξαναλέω, να δούμε τι γίνεται με τη διαχείριση των σκουπιδιών στις πόλεις, τι γίνεται με, ε, με την έρευνα σε αυτόν τον τομέα. Θα έπρεπε στα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν εκστρατείες και φόρουμ για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και να βρούμε τις καλύτερες λύσεις. Λύσεις που θα μπορούσαν να εγκρίνουν αργότερα οι περιφερειακές και τοπικές αρχές. Η Ευρώπη θέλει να παίξει αρχηγικό ρόλο στον αγώνα για τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο <coughs> και μόνο έτσι θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τα περιβαλλοντικά της προβλήματα η Ευρώπη. Το περιβάλλον θα το κληρονομήσουν τα παιδιά μας και δεν μπορεί η περιβαλλοντική πολιτική να ασκείται έτσι απομονωμένα, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες τις οι Πρέπει να δούμε τι γίνεται και με την βιομηχανία Χρειάζεται μία ενεργή και συνεκτική πολιτική περιβάλλοντος που να ανταποκρίνεται σε όλες τις προκλήσεις και σε οικονομικό επίπεδο. Χρειάζεται λογική χρήση των χημικών προϊόντων. Ήδη έχουμε εμείς έναν κατάλογο θα πρέπει βάσει αυτού του καταλόγου να απαγορεύσουμε τη, εντελώς τη χρήση όλων αυτών των ε, χημικών προϊόντων, να μετρήσουμε την τοξικότητά τους στο νερό, στις εκπομπές, στην κατανάλωση. Πρέπει να λάβουμε υπόψη την αηφόρο ανάπτυξη και όχι μόνο να σταθούμε στην πρόληψη από την ρήπανση. Η χημική βιομηχανία θα πρέπει στο, και στο μέλλον να μας εγγυάται μία λογική χρήση των προϊόντων με το μικρότερο δυνατό κόστος για το περιβάλλον. Θα πρέπει η Κομισιόν να επεξεργαστεί νομοθετικές πράξεις για αυτήν την αηφόρο χημεία. Εγώ στο έγγραφό μου προσπάθησα να αποδείξω την ανάγκη του να υποστηρίξουμε αυτό το πρόγραμμα. Ευχαριστώ τη Γραμματεία για τη δουλειά της. Ερμήνια, είσαι σκιώδης εισηγήτρια, έχεις το λόγο. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δουλειά της εισηγήτριας. Εγώ πιστεύω ότι πρόκειται για μια ολοκληρωμένη γνωμοδότηση, πρέπει να την υποστηρίξουμε πλήρως. Αδιαμφισβήτητα υπάρχουν δυνατότητες ε, να τροτοποποιήσουμε και να, την εμπλουτίσουμε την έκθεση η τοποθέτηση που μόλις ακούσαμε ε, μας ε, δείχνει ότι η συγγήτρια θέλησε να μας παρουσιάσει μία σύντομη πρώτη γνωμοδότηση για να μπορέσουμε όλοι να συνεισφέρουμε. Τώρα βέβαια ακούγοντας την προφορική παρουσίαση της εισηγήτριας πολλές από τις απορίες που είχα και λύθηκαν. Εγώ θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να, έχουμε, να διαμορφώσουμε μια διακλαδική, διατομεακή πολιτική για να παρεμβαίνουμε πιο ολοκληρωμένα στη χρήση των κονδυλίων για την πρόθεση των περιβαλλοντικών πολιτικών. Είναι επίσης σημαντικό να, σημαντική η αναφορά επέκτασης ε, της ε, συνεργασίας μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. όπως επίσης ε, και την ανάγκη που μας τόνισε η εισηγήτρια για την ανάπτυξη προληπτικών πολιτικών και αναφέρομαι σε δύο ζητήματα. Η μία αφορά την πρόταση της εισηγήτριας στο τέλος της πρώτης παραγράφου σχετικά με την ανάγκη νέων μέτρων για να αλλάξουμε την τροποποίηση προορισμού των εδαφών, κυρίως, ε, των γεών, κυρίως για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Εγώ νομίζω χρειάζεται μία εμβάθυνση, γιατί μία τόσο γενική προσέγγιση θα μπορούσε να είναι αποπροσανατολιστική. Θα ήθελα να ξέρω τι εννοούμε όταν μιλάμε για αλλαγή προορισμού. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η παραγωγή βιοκαυσίμων υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα η αλλαγή προορισμού των γεών θα πρέπει να, προστα... παρακολουθείτε για να μην έχουμε αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την αηφορία του. Το δεύτερο για τις νομοθετικές διατάξεις για την αηφόρο χημεία. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε. Προσθέτοντας πολλά από τα προφορικά επιχειρήματα της εισηγήτριας. Πρέπει να υποβάλουμε την πρόταση στην Κομισιόν. Σημερίζομαι την ανάγκη του να υπάρχει ένας ε, νομοθετικός ορισμός ε, για τη δράση της χημικής βιομηχανίας. Αλλά αυτή η αναφορά, χωρίς κανέναν άλλον προσδιορισμό, θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρερμηνίες και, παρεκ... και παρεκκλήσεις και στρεβλώσεις. <coughs> Πρέπει να τονίσω τη θετικότητα της αναφοράς που και στον τομέα των αποβλήτων Πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο η νομοθεσία για τα σκουπίδια. Υπάρχουν δυσκολίες στην επέκταση αυτής της ε, νομοθεσίας. και έχει ζητηθεί και στο παρελθόν γνωμοδότηση της Κομισιόν θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την ήδη και δουλειά. Θεωρώ λοιπόν ότι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ανακύκλωση των σκουπιδιών θα ήταν μια χρήσιμη δράση για την καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η γνωμοδότηση σε αυτή τη φάση διότι μας δίνει την δυνατότητα να αναλύσουμε το τι έχει γίνει στο παρελθόν για το έκτο πρόγραμμα. Να διαπιστώσουμε ποια λάθη έχουν γίνει. γιατί αρκετοί στόχοι δεν προσεγγίστηκαν. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το 7ο πρόγραμμα πιο ολοκληρωμένα, μειώνοντας ε, και τις πιθανότητες λάθους και αποτυχίες του προγράμματος του ιδίου. Ευχαριστώ η Κατρίν Φέρντερ για τους φιλελευθέρους. Ευχαριστώ και για την έκθεση και για τα σχόλια σχετικά με το κείμενο. Βέβαια, ήδη αναφερθήκαμε στην βιοποικιλότητα και στις ε, περιβαλλοντολογικές πολιτικές που ε, μας επηρεάζουν όλους γενικά σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε ε, σχετικά με ε, προβλήματα που φαίνονται πουσιώδη αλλά να αναθέσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση τη δυνατότητα να αναπτυχθεί και να τα επιλύσει και να σταματήσει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που διαπιστώνουμε στην Ευρώπη. Υπήρξαν ορισμένα σχόλια και πάντοτε είναι δύσκολα διότι περιοριζόμαστε ε, στο κείμενο που έχουμε ε, προς εξέταση γι' αυτό και θα προβώ σε ορισμένες τροπολογίες Ήδη όμως προηγουμένως αναφέρθηκα στον χώρο των πόλεων αλλά και της υπαίθρου και ο εισηγητής το ανέφερε. Πρέπει όμως να το πούμε σαφώς στην έκθεση αυτή. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο νομίζω ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Επίσης ο εισηγητής ε, μιλάει για τα απόβλητα αλλά ε, πρέπει να δούμε τη ε, διαχείριση των πόρων, την εξόριξη και τις αρχές που αναλαμβάνουν την επιτήρηση πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ διότι δεν σημαίνει μόνο ότι εξοριγνύουμε τους σπόρους αλλά συγχρόνως ρηπαίνουμε τους υδάτινους σπόρους και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν πρέπει να αποτελέσει βασικό στόχο του 7ου περιβαλλοντολογικού προγράμματος. Και το επόμενο θέμα επίσης αναφέρεται εδώ στις ανθρωπογενείς καταστροφές. Ε, πρέπει να βελτιώνουμε τις πολιτικές μας κατά τρόπον ώστε να φροντίζουμε οι φυσικές καταστροφές που πάντοτε συνέβαιναν όπως παραδείγματο χάρη οι σεισμοί και άλλα παρεμφερείς. Ε, βλέπουμε όμως ότι οφείλονται όλο και περισσότερο στους ανθρώπους με ε, αλλαγές του κλίματος, ε, με αλλαγές του ύψους των υδάτων, είναι δηλαδή διάφορα θέματα τα οποία πρέπει επίσης να εξετάσουμε και όσον αφορά την τελευταία παράγραφο εδώ μιλάμε για τα, ε, τις περιβαλλοντολογικές πολιτικές ε, και αυτό όπως συνήθως γίνεται ε, απλώς ένα ευχολόγιο, δηλαδή περιβαλλοντολογικός είναι ένας ωραίος όρος. Όταν όμως μιλάμε για πολιτικές πρέπει να μιλάμε για την απώλεια της βιοποικιλότητας, για τις κλιματολογικές αλλαγές, να αναρωτηθούμε ποια είναι τα προβλήματα και πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε και πώς δηλαδή ε, μπορούμε να, να στρέψουμε την διότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή την Επιτροπή. Προσβλέποντας προς το μέλλον πρέπει να πούμε ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους στόχους του 2020 και για την πολιτική συνοχή μετά το 2030 το, το 2030 θα πρέπει να μας απασχολήσει κατά τρόπον ώστε να δώσουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω των δράσεών μας τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν και να μειώσουν ότι το διοξίδιο του άνθρακος στην ατμόσφαιρα να έχουμε καλύτερες μορφές μεταφορών χρησιμοποιώντας τα κανάλια και επενδύοντας περισσότερο στα σιδηροδρομικά δίκτυα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλά στοιχεία και όπως όλοι οι συνάδελφοι προσβλέπω στις τροπολογίες και θα προβώ και εγώ σε ορισμένες. Ευχαριστώ όμως τον εισηγητή για την εξαιρετική αυτή έκθεση. Ε, ο Σον Πετρές δεν είναι εδώ, αλλά εσείς τον αντικαθιστάτε. Ναι, ναι, τον αντικαθίστω. Λοιπόν, εμείς ε, εκτιμούμε θετικά αυτή την έκθεση, δεχόμαστε τον συμβιβασμό με την ε, εισηγήτρια και θέλουμε να την βελτιώσουμε. Η περιβαλλοντική πολιτική είναι απόλυτα συμβατή με την πολιτική συνοχής. φορές στα σημεία 2 και 5 που ανέφερε η συγκήτρια σχετικά με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδίκησης είναι αυτές οι οποίες εφαρμόζουν την ε, περιβαλλοντική πολιτική ε, και είναι αυτές οι οποίες πρέπει να υλοποιήσουν τις εθνικές ε, ε, τις οδηγίες οι οποίες μεταφρόζονται σε εθνική νομοθεσία για παράδειγμα διαχείριση σκουπιδιών και του νερού που είναι και το πιο σημαντικό θέμα εμείς αξιολογούμε ιδιαίτερα θετικά το πλαίσιο να ανοίξουμε το 7ο πρόγραμμα με την διεύρυνση του δικτύου Natura 2000 και που είναι απόλυτα συνδεδεμένη και με τις πολιτικές συνοχής και δια της παρουσίας του ΦΕΝΤΕΡ. Θεωρούμε όμως αρκετά επικίνδυνη αυτή την ιδέα ε, αλλαγής προορισμού των ε, εδαφών, των γεών. Θεωρούμε ότι είναι κάτι το επικίνδυνο διότι θα μπορούσαμε τελικά σε περιοχές Natura να έχουμε να έχουμε πρόβλημα ως προς την εντατική γεωργία πρέπει να γίνει μια αναφορά για την βιοπικιλότητα θα πρέπει να το αναφέρουμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία και έχω το κείμενο και στη δικιά μου γλώσσα, πράγμα που ε, μου επιτρέψει να το κατανοήσω καλύτερα. Έχω δύο ερωτήσεις και ξέρω ότι εσείς θέλετε να έχετε σωστές ερωτήσεις. Στο σημείο 3, τι εννοούμε όταν μιλάμε για μία δίκαιη ισορροπία και αποφυγή νέων δαπανών. Γιατί εγώ υπήρξα δήμαρχος επί 15 χρόνια και θεωρούσα ότι οι επενδύσεις δεν είναι δαπάνες, είναι επενδύσεις ε, προς επίτευξη θέσεων εργασίας. Και ίσως το σημείο 5 ε, όταν έχουμε μια τέτοια γνωμοδότηση η οποία θα απευθύνεται σε μια άλλη επιτροπή η οποία είναι αρμόδια δεν θα έπρεπε να πούμε ότι για να ε, εφαρμοστεί η ε, περιβαλλοντολογική πολιτική χρειάζεται μια ισχυρή πολιτική συνοχής. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία παρατήρηση. Στην εισηγήτρια για το σημείο 3. όπου υπάρχει μία, ένας ορισμός μία, σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Πρόκειται για έναν τομέα που αφορά κυρίως την περιφερειακή πολιτική. Αυτή η προσαρμογή διότι οι κλιματικές αλλαγές που ε, διαπιστώνουμε σήμερα επηρεάζουν τομείς που αφορούν σε περιφερειακές οντότητες τύπου μεταφορές, γεωργία, τουρισμό κλπ. Και αυτό λέγεται σαφέστατα στην, έκθεση, στην αναφορά της Κομισιόν. Θα ήταν λοιπόν καλό να το πάρουμε και εμείς και να το βάλουμε στην έκθεση. Δεν έχω άλλους ομιλητές. Η κυρία Ντάντσικα. Ευχαριστώ για όλα σας τα σχόλια. Σχετικά με την αλλαγή του προορισμού των εδαφών. Εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα πρέπει να το τροποποιήσουμε, δεν πρέπει να αλλάξει. Χρειάζεται να έχουμε μία συγκεκριμένη αναφορά στα χημικά προϊόντα. Η χρήση τους ε, θα πρέπει να εμπλέκει τη χρήση νέων τεχνολογιών. Να έχουμε... να έχουμε μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση των χημικών. Τώρα για τα σκουπίδια χρειάζονται συγκεκριμένες προτάσεις σίγουρα και θα μπορούσαμε να έχουμε μία τροπολογία σχετικά. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή τον, τους συναδέλφους, τις προτάσεις τους, τις αμφιβολίες τους, τα προβλήματά τους. Μία έκθεση αυτού του στυλ έχει όρια, δεν μπορεί να είναι ιδιαίτερα μακροσκελής. Παρακαλώ να είστε σαφείς στις τροπολογίες σας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλό έγγραφο στο τέλος. 2 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι η κατάθεση τροπολογιών. Ολοκληρώνουμε. Ακούσαμε τις ε, βασικές ομάδες. Έχουμε ακόμη ένα σημείο στην ε, ημερήσια διάταξη που θα μπορούσαμε να τελειώνουμε γρήγορα, αλλά υπάρχουν προβλήματα μεταφοράς. Περιμένουμε τον Χόρστ Ράιχεμπαχ, ο οποίος είναι ο επικεφαλής της Task Force της ε, Κομισιόν, που θέσπισε πέρυσι η Κομισιόν και είναι υπεύθυνο για να βοηθήσει την Ελλάδα να αντεπεξέλθει από τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, ε, ε, πρόκληση και χρειάζεται ίσως να τον περιμένουμε λίγο. Παρακαλώ λοιπόν να ειδοποιήσετε ε, τους συναδέλφους σας στις πολιτικές ομάδες ότι καθυστερεί λίγο αυτή η συνεδρίαση για να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα στα πλαίσια του πακέτου λιτότητος και ανάπτυξης και ότι σύντομα θα ξεκινήσει η σχετική συνεδρίαση. Εν μεταξύ ατύπως διακόπτω τη συνεδρίαση. Δεν έχω όμως τη δυνατότητα να σας ειδοποιήσω, οπότε θα σας παρακαλούσα να παραμείνετε στα πέριξ. I would like also to tell you that we have sent the mail some minutes ago to all the entire committee to make people aware that it might be a little bit earlier than half past 11, so people should know. Μπορώ να ρωτήσω μία ερώτηση τον Πρόεδρο. Είπατε στις ανακοινώσεις ότι, στους συντονιστές ότι είχατε σοβαρές ε, αμφιβολίες. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν ποια είναι η αιτία των αμφιβολιών του Προέδρου. Ε, δεν ξέρω εάν πρέπει να υπάρξει μία κανονική αποστολή τριών ημερών ή αν πρέπει να είναι μία αποστολή εργασίας γιατί εδώ εκτός των συντονιστών έχουμε και τους, ε, ε, ε, τους εισηγητές που θέλουν να συζητήσουν στη Δανία με την Προεδρία αλλά και σαν Δανή με τους πολίτες της χώρας και ίσως δεν ε, πρέπει ε, να προσπαθήσουμε ε, να προχωρήσουμε. Είμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας. Οπότε όπως κάναμε και εις ε, την περίπτωση της Πολωνικής Προεδρίας ότι ε, δεν πρέπει να συζητούμε μόνο με τον υπεύθυνο Υπουργό για την ε, περιφερειακή πολιτική αλλά και με τους Υπουργούς Οικονομικών σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό και ανταλλαγή απόψεων για θέματα που μπορεί να επηρεάσουν το επόμενο τον επόμενο προϋπολογισμό. Οπότε ε, φαντάζομαι ότι θα πρέπει ε, να ε, βρεθούμε ε, σε θέση ανάμεσα εις ε, την συνεδρίαση του Απριλίου και του Ιουνίου να προετοιμαστούμε και να ε, χρησιμοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίδονται διότι ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή οι συζητήσεις για τον προπολογισμό δεν γίνονται σε επίπεδο υπουργών και πρωθυπουργών αλλά σε επίπεδο υψηλών στελεχών των Υπουργείων και φίλων της Προεδρίας οπότε ε, μπορούμε να κάνουμε να οργανώ... δεν ξέρω αν θα έχουμε ε, μία επικοδομητική ε, συνεδρίαση μαζί τους. Εγώ δεν ήξερα ποιος ήταν αυτός ο οποίος ήταν υπεύθυνος αλλά τώρα ξέρω. Ευχαριστώ. αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να καθίσετε, σας παρακαλώ. Ξεκινά η συνεδρίασή μας, οπότε ε, χαίρομαι πολύ που οι σοσιαλιστές με το ΕΛΚ συζητούν, αλλά θα παρακαλούσα τον συντονιστή σας να βρεθεί. Πού είναι ο συντονιστής σας? Λοιπόν, ξεκινάμε το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το οποίο θεωρούμε πολύ σημαντικό, διότι ο ρόλος μας της ε, πολιτικής ε, για να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να βοηθήσουμε την Ελλάδα να αναπτυχθεί είναι πολύ σημαντικό και θεωρούμε ότι πρέπει να συμβάλλουμε και να διευκολύνουμε ε, αυτή τη διαδικασία και να γι' αυτό προέβημαν στη γρήγορη ψήφιση του γενικού κανονισμού το φθινόπωρο αλλά θεωρούμε ότι και ό,τι θα βοηθήσει περαιτέρω στην Task Force και θα μπορέσει να οδηγήσει την Ελλάδα σε μία πρόοδο και την ελληνική οικονομία σε μία οδό ανάπτυξης θα πρέπει να επιβραβευτεί. Γι' αυτό και ζητήσαμε από τον κύριο Ράχενμπαχ εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έρθει εδώ και να μας παρουσιάσει τις απόψεις του. Θα θέλαμε επίσης να μας πει ε, ποιες είναι οι ανησυχίες του σχετικά με το τι άλλο χρειάζεται να γίνει και πώς διαβλέπετε τις ε, προοπτικές, δηλαδή αν υπάρχουν θετικές ε, ε, ενδείξεις στην Ελλάδα ότι κινείται προς ε, την ανάπτυξη ή αν βρίσκεται σε μία οδό η οποία χρειάζεται περισσότερες προσπάθειες για να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη. Τα σχόλιά σας θα μας είναι πολύτιμα και σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ευγνώμων για αυτή την πρόσκλησή σας να συζητήσουμε μαζί την κατάσταση της Ελλάδας και τις προπτικές όπως είπατε για περαιτέρω ανάπτυξη και για δημιουργία απασχόλησης και ιδίως για το ρόλο που μπορούν να παίξουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα μέτρα συνοχής. Όλοι γνωρίζουμε ότι τώρα είναι το πέμπτο έτος υφέσεως και μέχρι το τέλος της προηγουμένης χρονιάς υπήρχε μία επιτάχυνση της υφέσεως. Δεν νομίζω ότι το 2012 θα υπάρξει μία ανατροπή και δυνατότητα να επανέλθουμε σε μία πορεία αναπτυξιακή για την Ελλάδα αλλά ελπίζω ότι τουλάχιστον το 2012 θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για να τοποθετηθούν οι βάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Προφανώς το ε, ε, μακροοικονομικό πλαίσιο που καταρτίζει η Τρόικα και οι διαπραγματεύσεις για το PSI οι οποίες ε, συνεχίζονται και δεν έχουν καταλήξει είναι τα πιο βασικά στοιχεία για να δημιουργήσουμε μεγαλύτερη βεβαιότητα στην Ελλάδα διότι ε, ε, υπήρχε αυτή η φοβερή ανασφάλεια αν ε, και υπάρχει αν η Ελλάδα θα μπορέσει να καλύψει τις υποχρεώσεις της και να παραμείνει στο ευρώ και αυτή η ανασφάλεια εμποδίζει και την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις και εντός της Ελλάδος και από το εξωτερικό. Η κατάσταση είναι τέτοια ώστε ορισμένες επιχειρήσεις μεταφέρουν ε, τις έδρες τους εκτός Ελλάδος λόγω της δυσχερούς κατάστασης ε, από πλευράς πιστώσεων. Και αν υποθέσουμε, πράγμα το οποίο ακόμη είναι μεγάλη μπουκιά, ότι αυτά τα δύο ε, θέματα, το MOU και το PSI, τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν ε, ικανοποιητικά Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οποίες παραμένουν για την Ελλάδα στην προοπτική της ανάπτυξης που πρέπει να επιληθεί είναι ότι ο τραπεζικός τομέας της Ελλάδος αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στηρίξει την ε, οικονομία, αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της σοβαρής ε, ε, κρίσεως χρέους στην Ελλάδα και όχι διότι οι τράπεζες, τουλάχιστον η πλειοψηφία, οι μεγάλες τράπεζες, έχουν ε, κάνει ανόητες κινήσεις όπως άλλες, χώρες, ε, άλλες τράπεζες στην Ευρώπη. Ήταν σοβαρές τράπεζες όπως έχουν υποκαταστήματα στα Βαλκάνια και στην Τουρκία και ε, με την τάση όμως η οποία υπάρχει να διατηρούν ελληνικά ομόλογα έχουν τώρα πληγή και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν τις επιχειρήσεις και την ουσιαστική οικονομία. Για τον τομέα λοιπόν των επιχειρήσεων και τον ιδιωτικό τομέα στην Ελλάδα η στενότητα πόρων και πιστώσεων είναι μεγάλο πρόβλημα. Το άλλο σοβαρό θέμα είναι το επιχειρησιακό ε, πλαίσιο διότι βλέπετε ότι η Ελλάδα δεν έχει ένα καλό επιχειρησιακό περιβάλλον κάτι το οποίο δεν έχει άμεση σχέση με τα ταμεία συνοχής τα οποία διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά με τη δυνατότητα σωστής χρησιμοποίησεως αυτών των πόρων. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό η Task Force να μπορέσει να τονίσει και να επιλύσει το θέμα του ο επιχειρησιακού περιβάλλοντος, να μειώσει τη γραφειοκρατία, να απλοποιήσει τις εξαγωγές και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ένα από τα βασικά έργα στα, μέσω των οποίων θα μπορέσουμε να στηρίξουμε τις ελληνικές αρχές κατά τρόπον ώστε οι επιχειρήσεις και η Ελλάδα να γίνουν πιο θελκτικές, μάλλον οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα να γίνουν πιο θελκτικές. Και όσον αφορά τώρα το Ταμείο Συνοχής, αυτό καθεαυτό, έχουμε εργαστεί σε στενή συνεργασία με την ε, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακή περιφερειακής ε, πολιτικής, πολιτικής απασχόλησης, ε, την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα και με αυτές είχαμε ορισμένες επιτυχίες και μπορέσαμε να αλλάξουμε το ποσοστό συμμετοχής, πράγμα το οποίο οδήγησε σε καλύτερη αφομοίωση των διαρθρωτικών πόρων και ταμείων στην Ελλάδα και ήμασταν στο 33% στο τέλος του προηγουμένου έτους, πράγμα το οποίο δείχνει ότι υπήρχε μία βελτίωση και η αύξηση αυτή της αφομοιώσεως είναι ένας βασικός παράγων. Ενδεχομένως, ίσως γνωρίζετε ποια είναι τα μεγάλα προγράμματα. Υπάρχουν 100 οκτώ μεγάλα προγράμματα τα οποία παρακολουθούμε και των οποίων η πρόοδος ε, ε, παρακολουθείται και ελέγχεται αυτή ήταν η συζήτηση που είχαμε εχθές σχετικά με το μέσο συμμετοχής στον κίνδυνο που είναι πολύ σημαντικό κατά τρόπον ώστε ε, να επιλύσουμε το θέμα της χρηματοδότησης των υποδομών και τώρα θα έρθω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στη χρηματοδότησή τους. Υπάρχουν διάφορες δυνατότητες οι οποίες διατηρούν και που ε, έχουν συμφωνηθεί με τις ελληνικές τράπεζες. Το Aetian ε, ε, ε, συλλογικά δάνεια που έχουν προσυπογραφεί με αρμόδιες τράπεζες οπότε θα μπορούσε η Ευρώπη κάπως να στηρίξει τον και να υποκαταστήσει τον τομέα των ελληνικών τραπεζών αλλά επειδή όλα αυτά περνούν μέσα από τις τράπεζες οι τράπεζες δεν έχουν ρευστότητα δεν μπορούν να αναλάβουν περαιτέρω κινδύνους δεν καταβάλουν τα χρήματα χρήματα. Δεν πληρώνουν. Οπότε από αυτά τα πολύ σημαντικά και μεγάλα ποσά τα οποία έχουν διατεθεί ελάχιστα έχουν ε, διατεθεί και ε, αποδοθεί στην ελληνική οικονομία προσφάτως είχαμε μία συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ε, μία νέα δυνατότητα μέσω της οποίας η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει μισό δισεκατομμύριο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία θα, θα δανειοδοτήσει με ένα δις κατά τρόπον ώστε να συμβάλλει στην επίλυση της κρίσεως ρευστότητος που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές τράπεζες. Η ιδέα είναι ότι αυτή η δυνατότητα θα υπάρξει και θα υλοποιηθεί μέχρι το Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, οπότε οι τράπεζες τότε θα είναι καλά εξοπλισμένες για να μπορέσουν να προχωρήσουν διότι οι δυνατότητες ε, η δυνατότητα που θα δώσουν 2 ε, δισεκατομμύρια ευρώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουμε ε, το πρόγραμμα ανάπτυξης και εάν αυτό δεν επιτευχθεί οι μεγάλες δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν θα χαθούν. Αυτά ουσιαστικά είναι τα βασικά θέματα μαζί με την, ε, ε, ε, μαζί με τα θέματα που εξετάζουμε με τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η τράπεζα θα συμβάλλει αλλά και οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να συνεργαστούν και η προετοιμασία για να διατεθεί αυτό το ποσό όχι μόνο για χορηγήσεις επενδύσεων επενδύσεων αλλά και για κεφάλαιο κινήσεως θα πρέπει να διατεθεί και οι αποφάσεις έχουν ληφθεί μετά από την απόφαση της Επιτροπής των Κρατών Μελών. Οπότε, οι ανάγκη της Ελλάδας είναι πολύ μεγάλες. Οι δυνατότητες να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα είναι εξαιρετικές, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά εφέτος για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το δυναμικό. Το δεύτερο βασικό θέμα, το οποίο συζητήσαμε εχθές, και θα ήθελα να το ξανασυζητήσω σήμερα είναι οι παραχωρήσεις οι οποίες είναι ένα πολύ πολιτικοποιημένο θέμα δηλαδή μια ένα πολιτικό μήνυμα ότι τα πράγματα στην Ελλάδα προχωρούν και είναι αναγκαίο κατά τρόπον ώστε να είναι κανείς επισκεπ... Ε, ε, πιστευτός ε, και να δώσει το μήνυμα στον ελληνικό λαό ότι τα προγράμματα αυτά όντως συνεχίζουν να αναπτύσσονται είναι σημαντικά για την ανάπτυξη, είναι σημαντικά για την απασχόληση. Ε, έχουμε 10.000 ε, θέσεις εργασίας που εξαρτώνται από αυτά και ως εκ τούτου είμαι πάρα πολύ ευγνώμων διότι από όσο μπορώ να κρίνω από τη συζήτηση που είχαμε εχθές το Κοινοβούλιο στηρίζει πάρα πολύ ενεργά την προσπάθεια αυτή και ελπίζω ότι και στις συζητήσεις που θα έχουμε σήμερα το απόγευμα με τα κράτη-μέλη θα υπάρξει η αναγκαία στήριξη για την προσπάθεια αυτή. Το τελευταίο θέμα το οποίο θα ήθελα να αναφέρω διότι δείχνει πάρα πολύ καλά την ε, ε, αλληλεπίδραση που υπάρχει με ε, τα διαρθρωτικά ταμεία και ποιος είναι ο κίνδυνος για την Ελλάδα αν δεν υπάρχει ορθή χρήση των διαρθρωτικών ταμείων είναι η διαχείριση των αποβλήτων διότι υπάρχει μία διαδικασία για να κλείσουν οι χωματερές και να δημιουργήσουν νέα νέες εγκαταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει, να δημιουργήσει αυτές τις νέες θέσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων. Πιστεύουμε ότι τα πόροι θα βοηθήσουν και συζητούμε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να επιταχύνουμε και να προσφέρουμε την αναγκαία τεχνική βοήθεια ε, για τα τις προσπάθειες οι οποίες πρέπει να γίνουν σε αυτό το τομέα. Τελευταίο. Ποιες είναι οι δύο μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης τις οποίες έχουμε εντοπίσει μέσω μιας πολύ ενδιαφέρουσας μελέτης της εταιρείας McKenzie και η οποία πρέπει να ενδιαφέρει όλους αυτούς οι οποίοι ε, θέλουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της Ελλάδος. Σας συνιστώ λοιπόν ε, και μπορούμε να σας στείλουμε τη μελέτη αυτή. Οι δύο βασικοί τομείς αυτοί είναι αφενός η ενέργεια και συγκεκριμένα η ηλιακή ενέργεια και ο Υπουργός Περιβάλλοντος συνεργάζεται ε, στενά και πολύ σκληρά για να ε, μπορέσει να χρησιμοποιηθεί αυτή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ε, ενέργεια και να συμβάλλει στην ανάπτυξη μέσω του προγράμματος Ήλιος και έχει προχωρήσει μέχρι κάποιο σημείο. Το ερώτημα όμως είναι εάν πρόκειται για μία ευρία κλίμακα, εάν η ηλιακή ενέργεια θα έχει επαρκή ζήτηση και αν θα υπάρξουν συμβόλαια για εκμετάλλευση της ηλιακής ανεργίας, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει επιληθεί αλλά οι τεχνολογικές πτυχές είναι πολύ συγκεκριμένες και στην Ελλάδα η ηλιακή ενέργεια είναι σχεδόν ανταγωνιστική με τις παραδοσιακές πηγές ενεργείας. Άρα για την Ευρώπη αυτό είναι ένα μεγάλο συγκριτικό προτέρημα της Ελλάδος και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από την ευρωπαϊκή ε, οπτική γωνία. Το άλλο ήταν ο τουρισμός που πέρυσι πήγαινε καλά. Δηλαδή οι αμφιβολίες για την Ελλάδα βεβαίως σκιάζουν, επισκιάζουν και αυτό τον τομέα. Είναι ένας τομέας ο οποίος μπορεί να προβληθεί και ιδίως το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεως το οποίο περιλαμβάνει ε, κατά 50% ε, ακίνητο πλούτο θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί και να αναβαθμιστεί από την άποψη του τουρισμού. Υπάρχουν δυνατότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω των διαρθρωτικών ταμείων. Υπάρχει μία αναπτυξιακή προπτική για την Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να ξεκλειδωθεί εφέτος για να μπορέσουν να ξεμπλοκαριστεί, για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Πριν τώρα αρχίσουν οι ερωτήσεις και οι παρατηρήσεις από αυτόν, μήπως μπορείτε να μας δείτε δύο κουβέντες όσον αφορά την εντολή της Task Force. Πώς βλέπετε τον ρόλο σας τόσο ώστε να καταστούν τα πράγματα ξεκάθαρα, διότι ε, θεωρούμε ότι θα απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, αλλά για να το καταλάβουμε. Ράχινμπαχ. Η Task Force έχει διπλή εντολή. Πρώτα-πρώτα. Να παράσχει τεχνική άρρωγη στις ελληνικές αρχές, τόσο ώστε να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι για να μπορέσουν να πετύχουν τους διαφορετικούς στόχους που έχει θέσει η Τρόικα ε, όσον αφορά τις διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Να, επομένως, ποια είναι η βασική εντολή, γι' αυτό και μίλησα για το επιχειρηματικό περιβάλλον κλπ. Το άλλο κομμάτι της εντολής είναι το να βοηθήσουμε την Ελλάδα όσον αφορά την επιτάχυνση της συμμετοχής, της απορρόφησης των πόρων των διορθωτικών ταμείων με συνεργασία και σε συνεργασία με τις Γενικές Διευθύνσεις των διορθωτικών Ταμείων. Συνάδελφοι, πρέπει να σας ενημερώσω ότι εδώ έχουμε και τον ε, αναπληρωτή διευθυντή της ε, νομικής υπηρεσίας. Οπότε ε, μπορείτε να ρωτήσετε ό,τι ρωτήσετε. Γι' αυτό η Κράτσα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον επικεφαλής της Task Force, τον κύριο Ράμπραχτ, γιατί βρίσκεται σήμερα μαζί μας και μας δίνει απαντήσεις σε ένα θέμα το οποίο είναι βαθιά πολιτικό ε, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με πολλές τεχνητές και τεχνικές ε, διαστάσεις που αξίζει να τις αποσαφηνίσουμε. Εγώ ήθελα, καταλαβαίνετε ότι έχω επίγνωση αυτών των προκλήσεων και των προβλημάτων επειδή πρόκειται για τη χώρα μου. Ήθελα όμως να, ρωτήσω, να σας ρωτήσω κύριε Επικεφαλής ε, κάτι το στο οποίο αναφερθήκατε ήδη, ίσως θα ήταν ενδιαφέρον να μας εξηγήσετε περισσότερο, την ανάγκη κεφαλαίων κίνησης διότι οι διευκολύνσεις και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την οποία έχετε την επαφή και την επικοινωνία αφορούν την διευκόλυνση της εθνικής συμμετοχής για μεγάλα κομβικά έργα. Το κεφάλαιο κίνησης για μια οικονομία σε ύφεση που δεν καταφέρνει να αρχίσει την ανάκαμψη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπετε την καθημερινή κατάσταση των μικρών επιχειρήσεων που κλείνουν στη χώρα μου. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα, ένα θέμα που θέλω να θίξω και το άλλο. Η Ελλάδα και έχει ανάγκη και έχει δεσμευτεί να προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση. Ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η προετοιμασία ως προς το νομικό και το θεσμικό πλαίσιο για να μπορέσουν να γίνουν ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. I would ευχαριστώ. Λάμπερτ Φανίστερ, ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, κάθε μέρα μας έρχονται νέα μηνύματα από την Τρόικα σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης σε αυτή τη χώρα. Πρέπει να διαθέσουμε κονδύλια και πρέπει να έχουμε μία εικόνα πολύ πιο εμβαθυμένη για να ανοίξουμε νέες προπτικές. Ρωτώ. Πέρυσι πήγαμε η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στην περιοχή και τότε συνέπεψε η επίσκεψη με το ποσοστό συγχρηματοδότησης που δεν ήταν ιδιαίτερα ψηλό και είχαμε συζητήσει το πώς θα αλλάζαμε την κατάσταση. Πού βρισκόμαστε σήμερα. Αναφέρετε εσείς τις επενδύσεις, τις αηφόρες επενδύσεις, αλλά πώς μπορούμε εμείς να έχουμε εγγύησεις ε, ότι η επένδυση θα είναι η φόρα. Η κατάσταση είναι τέτοια σε αυτήν τη χώρα που δεν μπορεί κανείς να ξεκινάει με μια προϋπόθεση ότι όλα τα σχέδια είναι καλά. Τι γίνεται επίσης με την απορρόφηση σήμερα. Εσείς λέτε ότι οι χρηματικές ροές αφορούν στους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις, αλλά τι γίνεται ακριβώς με τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων. Υπάρχουν ακόμη δυσκολίες σχετικά. Αναφέρατε την ενέργεια. Είπατε ότι ο τομέας της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικός και χρειάζεται επενδύσεις. Και μιλήσατε για τους Κινέζους, μιλήσατε για δημοπρασίες. Μου φάνηκε ότι, αν κατάλαβα καλά, ότι γίνονται πολλές ε, μετατοπίσεις προς την Κίνα, επιχειρήσεων προς την Κίνα. ποιε είναι οι, χρηματο, οι χρηματικές ροές μεταξύ των δύο, δηλαδή με τους Κινέζους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θυμάμαι πολύ καλά ότι η πολιτική μου ομάδα είχε χαρεί πάρα πολύ ότι θα, θα πήγαινε αυτή η task force διότι θα μπορούσε να διατυπώσει προτάσεις για να υπάρξουν επενδύσεις, να ανακάμψει οικονομία και να μπορεί κανείς να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να κερδίσει χρήματα. Ήταν ίσως αφελές να πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο μπορούσε να γίνει ε, και όλα τα προβλήματα προβλήματα να λυθούν μέσα σε ένα τρίμηνο ή ένα εξάμηνο. Τα προβλήματα είναι πολύ δύσκολο για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να μπορούσαμε να έχουμε ε, μεταβιβάσει αυτή την ελπίδα καλύτερα. Πιστεύεστε ότι ε, στην Ελλάδα έχει γίνει αντιλεπτό ότι ε, δεν υπάρχει μόνο η επιταγή να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις αλλά και άλλα διότι δεν είναι μόνο προς συμφέρον της Ελλάδος να αντεπεξέλθει της κρίσης αλλά προς ολωνών ολονών μας και προσυμφέρον ολονών μας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ε, ατμόσφαιρα αισιοδοξία και προσμονής καλύτερου μέλλοντος για να ισχύσει κάτι τέτοιο. Διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το ότι πολλοί Έλληνες και πολλές επιχειρήσεις ε, ε, δεν, δεν σταθμίζουν έτσι τις δυνατότητες δυνατότητες τους γυρίζουν την πλάτη στη χώρα τους και αυτή, αυτό το έλλειμμα εμπιστοσύνης μου φαίνεται σαν ένα πολύ βασικό στοιχείο. Αυτό που θα με διέφερε να γνωρίζω και παρακολούθησε και χθε τη συζήτηση, δηλαδή δεν είναι σαφές αν τα κράτη-μέλη ε, ε, δεχθούν την, ε, την πρόταση αυτή για την αλλαγή του κανονισμού. Αλλά αυτό είναι πρόβλημα των κρατών μελών που πρέπει να επιληθεί σε επίπεδο κρατών και πρέπει να δούμε τι μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσει να στηρίξει την προσπάθεια μέσω μια σωστής εντολής. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα όντως να προχωρήσουμε ε, ε, σε μια πιο ορθόδοξο οδό διότι έτσι θα θέλαμε ε, να στηρίξουμε και να δείξουμε ότι στηρίζουμε την προσπάθεια για την Ελλάδα. Μπορείτε κύριε Ράχενμπαχ να ε, σχολιάσετε αυτά τα τρία θέματα. Ναι, σας ευχαριστώ. Όσον αφορά την ε, χρηματοδότηση αυτού του κεφαλαίου κίνησης, νομίζω ότι έχουμε μια σειρά μέσων σε σχέση με αυτό το startup. Άρα δεν λείπουν τα χρηματοδοτικά μέσα. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι το να δούμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα πλευρά των ε, τραπεζών να παράσχουν ε, τα χρήματα τα οποία χρειάζονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο δεν έχουμε μπορέσει μέχρι σήμερα να το επιλύσουμε. Τώρα, γενικότερα όσον αφορά τον ε, κλάδο επιχειρήσεων, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η υποστήριξη ε, σε σχέση με τις επενδύσεις δεν είναι τώρα το μέλλον το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η επιβίωση και πολλές τράπεζες κόψανε κονδύλια τα οποία έδιναν ακόμα και σε υγιείς επιχειρήσεις γιατί θα έπρεπε να συρρυκνώσουν τις εργασίες τους. Οπότε ακόμα και οι υγιείς επιχειρήσεις τώρα βρίσκονται ενώπιον δυσκολιών και αυτό το οποίο χρειάζονται είναι κεφάλαιο κίνησης. Επομένως, κάναμε την πρόταση και πήραμε το πράσινο φως τόσο ώστε και τα διαρθρωτικά ταμεία να μπορέσουν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση τώρα όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση ή τις ιδιωτικοποίησεις. Το ταμείο το οποίο θα πουλήσει τα ομόλογα, τα στοιχεία του ενεργητικού αυτά έχει ήδη συγκροτηθεί και έχουμε τώρα τρία είδη τέτοιων στοιχείων. Πρώτα-πρώτα έχουμε τις δημόσιες επιχειρήσεις που είναι το περίπου το 50% και για αυτές τις επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να υπάρξουν κάποιο είδους θεσμικά ή νομικά βήματα για να προετοιμάσουν την ιδιωτικοποίηση. Ακόμα δεν έχουν γίνει, οπότε έτσι θα προχωρήσει αυτό το μέτωπο και όσον αφορά τώρα τη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή τις ε, υποδομές, λιμάνια, ε, αεροδρόμια, έχουμε εδώ πέρα κάποια σειρά συγκεκριμένων μέτρων τα οποία πρέπει να γίνουν για να προετοιμάσουν την πώληση αυτών των ε, στοιχείων του ενεργητικού ούτω ώστε να προχωρήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και ο ελληνικός χώρος ιδιωτικοποίησης ε, ζήτησε τη στήριξη από τεχνικής για όλα αυτά. Τέλος, περίπου το 50% αυτών των στοιχείων ενεργητικού είναι γη ή ακίνητα. Αλλά τώρα είναι βέβαια θέμα κυριότητος του ακινήτου και είναι και θέμα επίσης χρήσης της γης επί των οποίων ο φορέας διωτικοποίησης έχει και αρμόδιτες που μπορούμε τώρα να επικαλεστούμε, τόσο ώστε σε σχέση και με το κτηματολόγιο ο μέλλον κύριος να έχει πραγματική κυριότητα. Και επομένω τώρα το θέμα είναι να είναι πιο αποτελεσματικό, πληρέστερο το κτηματολόγιο. Σε σχέση με αυτό, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική η δράση των Ολλανδικών αρχών και η συμπαράστασή τους. Όπως είπαμε, το θέμα της απορρόφησης και προφητικότητας από πλευρά της Ελλάδος είχαμε βελτίωση της επίδοσης αλλά ίσως εδώ ο ξαριστερών συνάδελφος θα ήθελε να σας τα πει όσον αφορά τώρα την εκροή των καταθέσεων αυτό είναι από τα μεγάλα προβλήματα που έχουν και αυτά και αυτό να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή ο ιδιωτικό ε, τομέα δεν έχει δείξει αλληλεγγύη όσον αφορά τη δύσκολη συγκυρία στη χώρα. Και αυτή η εκροή των καταθέσεων είναι πολλές δεκάδες δις λέγεται υπολογίζονται περίπου σε 50 δις αυτές οι ε, εκροές. Πάρα πολύ σημαντικό χτύπημα αυτό για τις ελληνικές τράπεζες. Για την Κίνα τώρα. Δεν είμαι σίγουρος ότι τι έχουν ακριβώς οι Κινέζοι. Είναι το θέμα αυτό του Λιμμένου στο Πειραιά έχει προχωρήσει η κατάσταση. Πάντως δεν έχουμε άλλες ε, πωλήσει αγορές από και προς τους Κινέζους. Τώρα να δούμε στον ενεργειακό τιμό τι τομέα τι έχουμε όσον αφορά τους μεγάλους παίκτες ε, οι οποίοι ενδεχομένω ενδιαφερθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε μία κατάσταση που συνολικά δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά συνεπάγεται και πολιτικά προβλήματα, να δώσει κανείς ένα μήνυμα ελπίδας. Και αυτό είναι που προσπαθώ. Κάθε φορά που βρίσκομαι στην Αθήνα, με περιορισμένα, περιορισμένη και επιτυχία και αξιοπιστία μέχρι στιγμής δυστυχώς. Διότι εάν κάποια στιγμή δεν υπάρξει μία μεταστροφή όπου οι άνθρωποι θα αρχίσουν να βλέπουν ότι κάτι αλλάζει προς το καλύτερο, τα μηνύματα αυτά δεν ε, μπορούν να στηριχθούν ε, δια των γεγονότων και φοβάμαι ότι αυτή η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα του συστήματος και η οικονομική ε, αβεβαιότητα ότι θα πετύχουμε το MU και το PSI μέσα στους δύο μήνες είναι μεγάλη και ε, ε, πολιτικά θεωρείται ότι αν αυτό επιτευχθεί θα έχουμε εκλογές ε, το δεύτερο ήμιση του Απριλίου ή του Μάιου πράγμα το οποίο εντείνει την αβεβαιότητα και υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν είναι εύκολο να εργαστούμε διότι αυτό το γνωρίζουμε και από άλλες περιοχές ότι η δυναμική και η προσπάθεια μειώνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά καταρχήν είμαι αισιόδοξο για το τι μπορούμε να πετύχουμε και για το τι τα κράτη-μέλη μπορούν να συμβάλλουν για την βελτίωση των δυνατοτήτων στην Ελλάδα. Ό,τι ε, υπάρχει είναι πολύ ενθαρρυντικό και δεύτερον, όπως έχω ήδη πει, είμαι της νόμης ότι για την Ευρώπη είναι πάρα πολύ βασικό σε μια τέτοια περίπτωση να μην αφήσει να καταρρεύσει η χώρα, αλλά να τη στηρίξει και οικονομικά και μέσω τεχνικής βοηθείας και μέσω των διαρθρωτικών ταμείων κατά τρόπον ώστε να υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον από αυτό το οποίο υπήρξε την τελευταία πενταετία. Τώρα, το ερώτημα εάν εδώ μπορεί να βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η πολιτική σας στήριξη για τις εργασίες και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο σύνολό της στην Ελλάδα και της Tax Force είναι ε, υψής της σημασίας. Και αυτή η πολιτική στήριξη θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στην ε, νομοθετική διαδικασία που έχει ξεκινήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσει να υλοποιηθεί και όπως είπα και χθε να τονίσουμε ότι αυτά μπορούν να βοηθήσουν και ελπίζω ότι τα κράτη-μέλη ε, θα ε, αξιολογήσουν με τον ίδιο τρόπο το νομοθετικό έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν και έχω ορισμένες επιφυλάξεις για την Ελλάδα όμως είναι ένα πολύ βασικό θέμα και ελπίζω ότι κάποια μέρα θα δουν το φως και τα κράτη-μέλη. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Εγώ θα ήθελα τώρα να σας πω κάτι όσον αφορά το επίπεδο απορρόφησης και όσον αφορά την κατάσταση για τα προγράμματα στατιστικές λένε ότι είμαστε στο 34,94% για την Ελλάδα όσον αφορά την απορρόφηση σε σχέση με το 33% που είναι ο μέσος κοινοτικό όρος. Τώρα ανοίξτε μια ματιά στο όσο προβλέπονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης. Είμαστε στο 39,65%. 34% είναι ο μέσος κοινοτικό όρος επομένως για το 2011 να κάνετε μια ανάλυση για τον στόχο του προπολογισμού οι στις πληρωμές έχουν πάει στο 104%. Αυτό σημαίνει ότι 2,6 δις ευρώ έχουν καταβληθεί στην Ελλάδα. Ένας άλλος τομέας τώρα, όπου εστιάζει την προσοχή μας πάρα πολύ, είναι το κλείσιμο του, των προγραμμάτων 2000-2006, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πέρσι καταφέραμε όλα τα προγράμματα του Ταμείου Ανάπτυξης να τα κλείσουμε. 27 που είναι πάρα πολύ αξιόλογη επίδοση και επομένω 581 ε, εκατομμύρια ευρώ καταβλήθηκαν για αυτό το λόγο επιπλέον στην Ελλάδα. Επίσης, άνοιξτε μια ματιά στην πραγματική κατάσταση, θα, θα διαπιστώσετε ότι η μεγαλύτερη απορρόφηση πέρσι οφείλεται στο ότι ο βαθμός συγχρηματοδότηση πήγε στο 85% και μετά συμπληρώθηκε με το 90%. 90% διότι καταφέραμε να κάνουμε τις τελικές καταβολές τον Δεκέμβριο σε αυτή την ε, συμπλήρωση. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό τον τόσο ψηλό στόχο και γι' αυτό και εστιάζουμε και συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην ποιότητα της ε, δαπάνης και εμείς και η Task Force. Και ακριβώς είναι πάρα πολύ σπουδαίος ο ρόλος της Task Force. Και συνεργαζόμαστε στενά με την Task για να δούμε ποιοι τομείς θα πρέπει άμεσα να μας απασχολήσουν και να δούμε τι γίνεται, τι, έχουμε πετύχει, τι μπορούμε να πετύχουμε στους προβληματικούς τομείς. Γι' αυτό και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα ε, απελευθερώσουμε τους πόρους ε, για τις μικρομεσαίες υπηρεσίες, όπως το είπε ο κ. Ράχιμπαχ, ναι, για τα κεφάλαια ε, κίνησης, όμως θα πρέπει να βρούμε τώρα και το κεφάλαιο εργασίας για να δούμε το πώς του χρόνου θα απελευθερωθούν αυτοί οι πόροι, θα φτάσουν στους τελικούς ε, ε, επιλέξιμους δικαιούχους και θα πρέπει επομένως να δούμε τι θα γίνει με την συγχρηματοδότηση, τι θα, πώς θα μπορέσουν να καταστούν εγγυητές οι τράπεζες, πώς θα μπορέσουν να βρουν τα σχετικά χρήματα για να δούμε και εμείς τι θα κάνουμε με τους δικούς μας πόρους. Βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί η η προσπάθεια για την απελευθέρωση των κλειστών ε, κλάδων, επαγγελμάτων κλπ. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για τα όσα πρέπει να γίνουν. Ε, ε, επομένως, πάρα πολύ σκληρά προσπαθήσαμε να δούμε ποια προγράμματα, ποια έργα θα κάνουν τη διαφορά. 181 τέτοια επισημάναμε σε αυτήν την λίστα. Ήδη τον Ιανουάριο θα γίνει αποστολή στην Ελλάδα για να εξασφαλίσουμε ότι η εποπτεία, η παρακολούθηση θα προχωρήσει για αυτά τα προγράμματα, αυτά τα έργα. Είμαστε αισιόδοξε. Γιατί έχουμε αμφιβολίες και ερωτηματικά για δύο-τρία μόνο από αυτά. Και ήδη έχουμε ε, διακρίνει για το εγγύς μέλλον κάποια ε, αποτελέσματα. Τώρα αυτά όσον αφορά την εφαρμογή και τώρα όσον αφορά την κατάσταση θα πρέπει να αναγνωριστεί τι γίνεται με τα μέσα του Ταμείου Συνοχής και την πολιτική συνοχής που είναι τα, πιο, τα μόνα πετυχημένα τώρα στην Ελλάδα. Οπότε ε, λέμε ότι έτσι θα παραμείνει προτεραιότητα η Ελλάδα καθοδόν προς την ανάπτυξη, προς την πάυση της κρίσης. Οπότε αυτά και για τη σημασία της τάξης φοράς. Γιώργος Σταυρακάκης και άλλοι δύο έχουν το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Χόρστ Ράιχνμπαρ και το επιτελείο του για όλες αυτές τις ε, απόπειρε να προσφέρει αρρωγή στην οικονομία τους ε, για αυτή την τόσο σημαντική γνωστή τεχνική που σε πολλούς τομείς μας προσφέρεται. Τα ξέρετε τώρα εδώ καιρό είπατε στην Ελλάδα. Έχετε λοιπόν εις βάθος γνώση της κατάστασης ελληνικής οικονομίας. Σας παρακαλώ, πέστε μας δύο λόγια παραπάνω όσον αφορά το νέο μέσο, αυτό το risk sharing management, αυτή την διαχείριση ε, επιμερισμού του κινδύνου. Πέτρο Ζήμαν. Κύριε Ράχεμπανκ, ευχαριστώ για τα λόγια σας. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πρώτο μέρος της εντολής σας και σε αυτό θα θέσω την ερώτησή μου, διότι ε, ε, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για προϋπόθεση για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το κράτος και το σύνολο. Η Task Force στο σημείο αυτό έχει ε, όπως είπατε σήμερα αλλά και στο παρελθόν αναλάβει διάφορα μέτρα τα οποία εφαρμόζει στα επίπεδα του εθνικού κράτους αλλά που είχα κάνει αυτή την ερώτηση και στην προηγούμενη συνάντηση και θα ήθελα απλώς μία ενημέρωση διότι ε, ε, είναι μία χώρα η οποία δεν έχει κάνει ποτέ μεταρρυθμίσεις στην διοίκηση από πάνω προς τα κάτω αυτό και δεν είναι δυνατόν εάν στην κορυφή δεν υπάρξουν αλλαγές να λειτουργήσουν ε, ε, στη βάση. Μπορεί να λειτουργούν στις, ε, στις, στη βάση σε μικρά γραφεία στην περιφέρεια. Αλλά τι δέσμευση έχει αποσπάσει η Task Force ή τι δυνατότητες διαβλέπει η Task Force εκτός από το top-down να να υπάρξει και μία εφαρμογή bottom-up, δηλαδή από κάτω προς τα πάνω, κατά τρόπον ώστε να υπάρξει η, η αντίστοιχη στήριξη εις, ε, της ε, πρώτου επίπεδου ε, αρχές, στη βάση δηλαδή και στο μεσαίο επίπεδο, κατά τρόπον ότι αποφασίζεται στην κορυφή να μπορεί να εφαρμόζεται μέχρι τη βάση. Κύριε Ράχιμπαχ, εκτιμώ πως έχετε αντιληφθεί αυτό το διάστημα εκτιμώ πως έχετε αντιληφθεί καλύτερα από άλλους την κατάσταση στην ε, χώρα μου. Από άλλους οι οποίοι υποστηρίζουν πολιτικές τιμωρίες και επιθαρχίες. Έχω σημειώσει ότι έχετε πει τρεις φορές ότι οι Έλληνες δεν μπορούν να σηκώσουν άλλα βάρη. Θα ήθελα να μου πείτε πώς εκφράζεται αυτό στην πολιτική που προωθείται. Ένα δεύτερο ερώτημα. Στην τριμηνιαία έκθεση της Task Force για την Ελλάδα γίνεται εκτενής αναφορά στην προώθηση της υλοποίησης μεγάλων έργων προτεραιότητας όπως τα πέντε μεγάλα έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων. Είναι σαφές ότι στόχος είναι η προώθηση της απορροφητικότητας των πόρων. Μιλήσατε στην αρχή και για 10.000 θέσεις εργασίας που θα προσφέρουν. Υπάρχουν όμως κάποια ερωτήματα. Υπάρχει προβληματισμός για το ποια θα είναι η κατεύθυνση της ανάπτυξης που επιδιώκεται. Αν για παράδειγμα επιστρέφει η χώρα στη λογική των αποσπασματικών μεγάλων έργων υποδομής του παρελθόντος και αν με τις επιλογές αυτές βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητά τη Επιπλέον, γιατί προκρίνεται η χρηματοδότηση τέτοιων οδικών έργων μεγάλων στο μέσο της κρίσης όταν στην Ελλάδα η χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου μειώνεται λόγω του υψηλού κόστους των καυσίμων και των διοδίων. Δεν κυκλοφορούν πια τα αυτοκίνητα. Και αντιθέτως εγκαταλείπεται ο σιδηρόδρομος. Η πολιτική της Τρόικας στην Ελλάδα καταργεί τα δύο τρίτα των σιδηροδρομικών γραμμών κάτι που είναι αντίθετο και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μια και έχει χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκά κονδύλια. Τώρα μην πω για το σιδηρόδρομο, έχει σαφώς μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, είναι πιο προσιτό στους οικονομικά αδύνατους και είναι όχημα ανάπτυξης για μας για τον 21ο αιώνα. Το τρίτο ερώτημα είναι ποια θα είναι ακριβώς η ανάμειξη της Task Force στο σχεδιασμό της πολιτικής συνοχής για την Ελλάδα μετά το 2013 και ποια άποψη έχει για το περιεχόμενο της πολιτικής αυτής για τη χώρα στο μέλλον. Και το τέταρτο ερώτημα είναι σχετικά με την αυτοδιοίκηση, μια και αναφέρεται στην έκθεση ότι είναι θετική η πρόσφατη μεταρρύθμιση που εμείς το λέμε καλή κράτη. Πώς θα ενισχυθεί η αυτοδιοίκηση στο ρόλο της για την ενδογενή τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής συνοχής όχι μόνο μέσα από τα μεγάλα έργα αλλά και μέσα από σχέδια σε τοπική περιφερειακή κλίμακα. Και με την ευκαιρία, αν μπορούσατε να ξεκαθαρίσετε τις διαφορές των ρόλων με τον κύριο Φούχτελ που έχει, από ό,τι διαβάζουμε, εστιάσει στο θέμα της αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει ο Θα προσπαθήσω να σας ε, εξηγήσω ακόμη μια φορά την ε, σημασία αυτού του μέσου επιμερισμού του κινδύνου. Όπως προανέφερα, οι τράπεζες σήμερα δεν προτίθενται πλέον να αναλάβουν περαιτέρω κίνδυνο για την Ελλάδα, δεν έχουν τη ρευστότητα, δεν μπορούν να βοηθήσουν επομένω την ε, εκτέλεση συγκεκριμένων προγραμμάτων και έργων και συγκεκριμένα όσον αφορά τον τομέα των υποδομών. Αυτό ε, έχει, έχει αποτελέσει τεράστια τροχοπέδη διότι χρειάζεστε μακρόπνοη χρηματοδότηση για αυτά τα έργα της υποδομής. Χωρίς αυτή τη χρηματοδότηση δεν είναι δυνατόν να έχετε ανάπτυξη τέτοιων έργων και προγραμμάτων επομένως. Η ουσία αυτού του μέσου είναι το να μπορέσει να εξεύρει κάποιες δυνατότητες για τις τράπεζες. Και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η υπόθεση των υποδομών. Και έτσι να ξεκινήσουν ή να ολοκληρωθούν όσοι έχουν ξεκινήσει από αυτά τα έργα και προγράμματα Οπότε και ερχόμαστε στην ε, ερώτηση. Τι έγινε με αυτές τις εκχωρήσεις, παραχωρήσεις, τις προβλέψεις για την απελευθέρωση. Που φυσικά όλα αυτά τα έχει φρενάρει κρίση. Το θέμα είναι τώρα τι θα γίνει με το, το, αν θα ξεκινήσουν ή όχι αυτά τα έργα. Το θέμα είναι επίση αν, αν θέλει κανεί να ολοκληρώσει, να τελειώσει τα σχετικά έργα, διότι υπάρχουν συμβάσεις μεταξύ ε, ε, των, του κράτους και των εταιριών, μεγάλες εταιρείε από Ισπανία, Γερμανία και Γαλλία, που φυσικά και έχουν πάρα πολύ σημαντικές αξιώσεις κατά του ελληνικού δημοσίου, εάν αφαιτηθούν οι συμβάσεις και δεν συνεχιστούν τα έργα, επομένως. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο λοιπόν θα, θα, θα κοπούν τα έργα, θα σταματήσουν και χρησιμοποιηθούν αλλού τα χρήματα. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχουν αυτέ οι τεράστιε γιγαντιέ αξιώσει εάν δεν ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Και... Άρα πρέπει να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και άλλωστε υπάρχει και συμβολική αξία και σημασία για το μέλλον τη Ελλάδος. Είναι αυτό. Άρα ολοκλήρωση, αποπεράτωση και επομένως με το μέσο επιμέρισμα του κινδύνου έχουμε τώρα εδώ πέρα ένα κρίσιμο κομμάτι στο ψηφιδωτό και βέβαια χρειάζεται συνδυασμένη προσπάθεια ούτως ώστε να γίνει αυτή, αυτή η φάση. Υπήρξαν και δύο ερωτήσεις σχετικά με την ανάγκη όχι μόνο να προσπαθήσει κανείς να προβεί σε μεταρρυθμίσεις επικεντρικού επίπεδου αλλά και επί περιφερειακού και τοπικού επίπεδου το οποίο ίσως δεν, είναι, δεν υπήρξε η πρώτη προτεραιότητα και ακριβώς ε, για αυτήν την πτυχή της ε, μεταρρυθμίσεως της δικήσεως ε, δεν είχαμε τόσες δεν είχαμε ούτε μία σαφή εικόνα ούτε έναν αριθμό συστάσεων από τον ΩΣΑ από την έκθεση την οποία φαντάζομαι όλοι γνωρίζετε είναι όμως σίγουρα ένας τομέας που είναι πολύ σημαντικός και ο οποίος έχει συζητηθεί με τον Υπουργό Εσωτερικών που είναι υπεύθυνος για το θέμα αυτό. Δηλαδή ε, ε, αυτός είναι υπεύθυνος στο Κεντρικό ε, Υπουργικό Συμβούλιο για την εσωτερική ρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και συγχρόνως και με την τοπική αυτοδιοίκηση η οποία πρέπει να ενισχυθεί κατά τρόπον ώστε τα προγράμματα να μπορούν επίσης να εφαρμόζονται στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και άλλα βασικά θέματα που προανέφερα όπως η διοίκηση των αποβλήτων να τη χάνουν μιας καλύτερης διαχείρισης. Όσον αφορά τον ρόλο του συγκεκριμένου μηχανισμού για την Ελλάδα έχει αναλυφθεί από την Γερμανία και η Γερμανία έχει αναλάβει να συζητήσει από κοινού με τις ελληνικές αρχές αλλά και με την τοπική αυτοδιοίκηση κατά τρόπον ώστε να καταρτιστεί ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί υπό την κατεύθυνση των γερμανικών αρχών. Η έχει δραστηριοποιηθεί στο τομέα αυτό και αυτή τη στιγμή έχουμε τουλάχιστον μία κίνηση των εργασιών ε, οι οποίες είναι στο σωστό δρόμο για να μπορέσουν να καταλήξουν. Δεν είμαι εις θέση να σας ε, περιγράψω με ακρίβεια τον ρόλο του κυρίου Φούχτελ, οπότε όμως γνωρίζω. Υπάρχει ένας ε, φορέας, ομάδα, όπου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, τέλο πάντων ρωτήστε εκείνον καλύτερα. Τώρα, όσον αφορά του σιδηροδρόμου, ίσω υπάρχει εδώ συνάδελφο η οποία Γνωρίζετε σχετικά και μπορεί να πει δύο λόγια διότι και εκείνη συμμετέσχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα θέματα μεταφορών. Έχει μακρά θητεία, οπότε μπορεί να σας τα πει καλύτερα. Όσον αφορά το μέλλον της πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα. Βεβαίω και είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα και συγκεκριμένα. Έχουμε την Γενική Διεύθυνση για την Περιφερειακή Πολιτική και όπου οι ε, ελληνικές αρχές θα πρέπει να προβούν στις αναγκαίες ε, προετοιμασίες. Πάντως, θα πρέπει να τονίσω το ότι προσπαθούμε να βοηθήσουμε την Ελλάδα να εφαρμόσει τα σχετικά, διότι υπάρχουν πολλές ιδέες, υπάρχουν προγράμματα δράσης αξιόλογα, υπάρχουν ε, προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης. Αυτό το οποίο όμως εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι όλα αυτά να υλοποιηθούν, όλα αυτά να γίνουν πράξη στην πραγματική οικονομία. όπως προβλέπετε. Ευχαριστώ πολύ. Διευθυντά. Αν δούμε περιφερειακό και κεντρικό, αν δείτε τη διαχείριση των ε, διευθυντικών ταμείων, θα διαπιστώσετε ότι έχουμε πέντε εθνικά και πέντε περιφερειακά προγράμματα. Επομένως, δουλεύουμε και σε επίπεδο περιφερειών και αυτό πάει να πει ότι η διαχείριση γίνεται σε περιφερειακό επίπεδο. Ε, ο Επίτροπος είχαν εμπιστευτεί την χώρα, είδε τους εκπροσώπους των περιφερειών και με δεδομένα αυτά τα προγράμματα έχουμε και ε, κάποιο είδου ε, τεχνική αρρωγή, ούτως ώστε μπορούν να προωθήσουν καλύτερα οι τοπικές αρχές τα κονδύλια συνεχώς έχουμε και αναθεώρηση αυτής της ε, αρρωγής τόσο ώστε να μπορούμε να πλαισιώσουμε καλύτερα τις σημερινές ανάγκες και εάν τώρα ρίξετε μία ματιά στα βασικά έργα, έχουμε τα 181, δεν, δεν είναι όλα το ίδιο σημαντικά, υπάρχουν μερικά τεράστια έργα ε, και ε, όπως είπε ο Γιώργο Ράχινμπαχ, είναι πάρα πολύ σημαντικά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεωρήσει ότι είναι έργα ευρωπαϊκής προσθεμένης αξίας. Επομένως είπαμε ότι υπάρχουν και κάποια άλλα έργα τα οποία είναι έργα γέφυρες και άρα και αυτά επίσης δεν είναι δυνατόν να αφαιθούν αν ολοκληρωτά. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος αν δεν τελειώσουν. Όμως θα πρέπει να γίνει η διόρθωση της προηγούμενης περίοδου. Είναι, πάρα, πάρα πολύ σημαντικέ οι οικονομικές επιπτώσεις για το ελληνικό κράτος. Επομένως, μέσα σε αυτά τα 181 έργα, τα οποία περιέχονται στα ε, επιχειρησιακά προγράμματα, είναι εκτός από τα μεγάλα, έχουμε και κάποια μικρά έργα και στο επίπεδο εκείνων των μικρότερων έργων συνεργαζόμαστε και με τις περιφερειακές αρχές. για τους σιδηρόδρομους. Αθήνα Πάτρα, Αθήνα Σαλονίκη, οι συνδρομικές γραμμές έχουν αναβαθμιστεί ε, και, και αυτό είναι μέσα στα 181 έργα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αποσπάσει έναν ειδικό όσον αφορά τις ε, υποδομές ε, στα έργα μεταφοράς και ο συνέδρος αυτό συνεργάζεται με τις εθνικές αρχές, με την ε, Γενική Διεύθυνση για τα Περιφερειακά, με εμά, ε, ε, ω έργο έτσι του αρμόδιου φορεί, ούτω ώστε να τα καταφέρουν να υλοποιήσουν ό,τι προβλέπεται. Επομένω, και εμεί προχωρούμε να δούμε τι γίνεται με το βαθμό ρημότητα, με το βαθμό υλο... δυνατότητα υλοποίηση του προγράμματο. Και αυτά λοιπόν τα έργα για του δρόμου περιέχονται στα 181 και επομένω σε κάποια φάση πρόκειται να ολοκληρωθούν. I would Σας ευχαριστούμε και ολοκληρώσαμε σε αυτό το σημείο και από ό,τι γνωρίζω. Και κατάλαβα πολλά έχουν γίνει, όμως ακόμη θα πρέπει να γίνουν και άλλα και γι' αυτό και θεωρούμε εδώ στο Κοινοβούλιο ότι είναι αυτό το οποίο είπε η Κωνσταντζα, το τι μπορούμε να κάνουμε. να προχωρήσουμε με αυτό το μέσο της, του εμμερισμού του κινδύνου όσο είναι πιο γρήγορα. Θα πρέπει βέβαια συνάδελφοι και η Ελλάδα να προετοιμαστεί για το αύριο. Είναι αυτό ξεκάθαρο. Επομένω ελπίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτή θα το λάβει αυτό υπόψη. Το τι θα γίνει και αύριο, γιατί πρέπει να συνεχιστούν όλα αυτά τα έργα. Και πάλι σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Και καλή επιτυχία στο έργο σας που τόσο χρησιμοποιεί για την Ελλάδα. Πέρασε η Ανδριάσου, θα τα ξαναπούμε τέλος Φεβρουαρίου, δεν θυμάμαι ποια μέρα.